Good afternoon everybody. We are running a bit late already. Καλησπέρα σας. Έχουμε κάπως καθυστερήσει. Έρχονται σιγά σιγά οι συνάδελφοι και οι υπεύθυνοι του τμήματος πολιτικής, οπότε νομίζω ότι μπορούμε να αρχίσουμε και θα ήθελα να αναφερθώ στις αποφάσεις των συντονιστών σήμερα το πρωί. Η έγκληση της ημερήσιας διάταξης για την 3η Δεκεμβρίου έγινε δεκτή με κάποιες αλλαγές. Χρειάζεται να πω τους αριθμούς. 2214 και 2449 του 2015 που ζήτησε το ΕΛΚ θα συμπεριληφθούν στην ημερήσια διάταξη τον Ιανουάριο ή αργότερα. Οι 1062 και πολλές ε, αναφορές για την ηλιακή ενέργεια που ζήτησε η ΓΚΟΕ θα ε, συμπεριληφθούν ε, στην ημερήσια διάταξη του Φεβρουαρίου του 2016 και λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι η μελέτη του Τμήματος Πολιτικής θα είναι έτοιμη το Φεβρουάριο, η 1956 του 2012 και άλλες αναφορές για το ίδιο θέμα που επίσης ζήτησε η ΓΚΟΕ θα συμπεριληφθούν στην ημερήσια διάταξη του Δεκεμβρίου οι συντονιστές αποφάσισαν για τη διαδικασία, την προφορική ερώτηση για τα, ε, παιδικά, για τα δικαιώματα των παιδιών ε, και αποφάσισαν να συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη του Δεκεμβρίου. Δεύτερον, η γνωμοδότηση για την έκθεση ε, Γιούρι όσον αφορά την παρακολούθηση του, της ενωσιακής νομοθεσίας, ε, ετήσια έκθεση, θα γίνει βάση της διαδικασίας ΔΕΟΝΤ. Ε, θα επανέλθουν αργότερα για να μας πούν κατά πόσο θέλουν ή όχι να την αναλάβουν. Αν όχι, εγώ ως πρόεδρος έχω ε, ε, αποφασίσει να την κάνω η αναφορά 052 του 2015 για την ε, καταπολέμηση της υπατήτητας γάμα. Θέλουμε να συμπεριληφθεί στην μερίσια διάταξή μας αυτή τη στιγμή μας απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά πάσα πιθανότητα Φεβρουάριο ή Μάρτιο. Τώρα, όσον αφορά τώρα τις επίμαχες αναφορές, συμβιβαστικές ε, λύσεις ε, που πρότεινα έγιναν δεκτές για διάφορες αναφορές, η συμβιβαστική λύση που πρότεινα ενέκρινε κάπως τροπο, ενεκρίθη κάπως τροποποιημένη για την 2635 του 2014 και την 89 του 2015. Οι συντονιστές αποφάσισαν ότι στην περίπτωση της αναφοράς 0052 του 2015 η μελέτη η οποία έγινε το 2012 θα αποσταλεί στον αναφέροντα και ο αναφέρον Επίσης ε, θα λάβει τη σύσταση να ε, απευθυνθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Εν τω μεταξύ θα αποσταλεί επιστολή και από εμά στη μόνιμη αντιπροσωπεία για να ζητηθούν περαιτέρω διευκρινήσεις και θα παραμείνει ανοιχτή η αναφορά μέχρι την απάντηση της Ρουμανικής Μόνιμης Αντιπροσωπείας ε, σε μας, στην Επιτροπή μας. Οι συντονιστές αποφάσισαν ε, την αναφορά 0074 του 2015 να τη διατηρήσουν ανοιχτή μέχρι την ολοκλήρωση της γνωμοδότησής μας ε, για το UNCRPD και το αίτημα της ε, ΓΚΟΕ έγινε δεκτό για την 2164 του 2014. Έτσι λοιπόν πράξαμε για τις επίμαχες αναφορές, ήμασταν πάρα πολύ αποτελεσματικοί και με πάρα πολύ, με επαγγελματικό τρόπο λειτουργήσαμε όσον αφορά την πύλη, τη διαδικτυακή της επιτρέπουν αποσταλεί κάποια έγγραφα σχετικά. Η διερευνητική αποστολή που θα λάβει χώρα από τις 8 στις 10 Φεβρουαρίου του 16 στην Ισπανία κατά τη διάρκεια της πράσινης εβδομάδας εν ολίγης. Ε, το πρόγραμμά της θα αποφασιστεί το Δεκέμβριο και οι συντονιστές θα πρέπει να μας γνωστοποιήσουν ε, τα ονόματα των ε, ενδιαφερομένων μελών στη γραμματεία της Επιτροπής μας μέχρι τις 26 Νοεμβρίου. Θα γίνει δημόσια ακρόαση λαμβάνοντας υπόψη τα, ανησυχίε των πολιτών μας βάσει του άρθρου 51. Οι συντονιστές θα προτείνουν ενδεχό, ε, θα προτείνουν κάποιους υποψήφιους ομιλητές και θέματα προς συζήτηση πριν από τις 20 Νοεμβρίου. Μένουν ακόμη μερικές μέρες. Όσον αφορά την προφορική ερώτηση ή ψήφισμα για τη συνθήκη του Μαρακέφ, είναι ένα θέμα που χρόνια ε, τίθεται. Και επειδή η Γιούρη Νομοθετική Επιτροπή επ' αυτού αποφασίσαμε ότι θα, θα αναζητήσουμε μια συμφωνία μαζί τους για το πώς να προχωρήσουμε. Από ό,τι καταλάβαμε από τους συντονιστές ε, που έγνεφαν καταφατικά, ε, θέλουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ορατότητα για το θέμα αυτό. Αν γίνεται να υπάρξει μια προφορική ερώτηση, ένα πλήρες ψήφισμα όλο με ε, συζήτηση στην Ολομέλεια, προκειμένου και ψηφοφορία ε, για να πιεστούν τα κράτη-μέλη να επικυρώσουν ε, τη συνθήκη. Είναι κάτι το οποίο βέβαια πρέπει να εγκριθεί από τη διάσκεψη των Προέδρων και αν δεν γίνει κάτι τέτοιο έχουμε μια θέση αναδίπλωσης η οποία θα είναι να περιοριστούμε σε ένα σύντομο ψήφισμα το οποίο δεν ε, συμπεριλαμβάνει απαραίτητος συζήτηση στην Ολομέλεια, συμπεριλαμβάνει όμως ψηφοφορία. Αυτά λοιπόν αποφασίσαμε. Ως προς το ερευνητικό μας πρόγραμμα, οι συντονιστές έλαβαν γνώση των σχετικών προτάσεων. 19 Νοεμβρίου είναι η προθεσμία για την κατάθεση περαιτέρω προτάσεων. Θα εγκρίνουμε το πλήρες πρόγραμμα στην επόμενη συνεδρίασή μας το Δεκέμβρη. Επίσης αποφασίσαμε να ζητήσουμε δύο μελέτες από το Τμήμα Πολιτικής. Πρώτον για την υποστήριξη της ε, ακρόαση του Φεβρουαρίου για τα ε, θεμελιώδη δικαιώματα και δεύτερον για ε, τη συνθήκη του Μαρακές για να τονίσουμε και πάλι τη σημασία ε, του ψηφίσματος. Όσον αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές, έκανα έκκληση στους συντονιστές να λάβουν γνώση της ε, δέσμευσης τη Επιτροπής να το ολοκληρώσουμε μέχρι τα τέλη του έτους, που έχει αρχίσει μια εργασία που έχει αρχίσει εδώ και πάνω από έξι μήνες ε, και έχει κρατήσει πολύ αυτή η διαδικασία, αν σκεφτεί κανείς ότι είναι μια διαδικασία λειτουργίας εσωτερικής δική μας και όχι αναφορές των πολιτών, πρέπει να τη διαχειριστούμε με πολύ καλό και επαγγελματικό τρόπο και να είμαστε κατά το μέγιστο αποτελεσματικοί ενημερωτικά πολλά ε, σημεία ε, ήταν ενημερωτικά ε, ένας μεγάλος, μακρύς κατάλογος θεμάτων και υπάρχουν άλλα τρία τα οποία θα εγγραφούν στο κατάλογό μας προς ενημέρωση για το Δεκέμβριο. Αυτά λοιπόν από τους συντονιστές. Τώρα νομίζω ότι έφτασε η ώρα να περάσουμε στις αναφορές μας. Και χαίρομαι που καλωσορίζω σήμερα τον Άφεν Πράντε και τον κύριο Χίλτε, όσον αφορά την αναφορά 2482 του 2014 όσον αφορά την αεροπλοεία και το πώς μπορούμε να τη δαμάσουμε τα, το θόρυβο των αεροσκαφών ε, από ε, την πολιτική αεροπορία όσον αφορά ε, την προτινόμενη απαγόρευση των νυχτερινών πτήσεων και την κατάργηση των φορολογικών προνομίων της αεροπορικής βιομηχανίας. Επίσης αναφορά υπαριθμών 2664-2014 του Μάνφερ Πράντε, δαμάζοντας την αεροπορία και ναι. πάλι με συγκεκριμένη αναφορά στο θόρυβο από νυχτερινές πτήσεις στον αερολιμένα κολονίας Βόνης και αναφορά 2670 του 2014 της Πέτρα Χέπτενμάχερ για το θόρυβο των αεροσκαφών από τον αερολιμένα Κολονίας και και πάλι. Θα ήθελα λοιπόν τώρα να σας δώσω το λόγο. Ε, Σουζάν Γέγκερ, Μάνφρεντ Πράντε, έχετε το λόγο για 5 λεπτά. Okay. Thank you for being allowed to make σας ευχαριστώ που μας επιτρέπετε να κάνουμε μια δήλωση. Λέγομαι Χέγκερ, είμαι από την Αυστρία. Είμαι μία από τις δύο που πήραν την πρωτοβουλία για το λεγόμενο taming avia. Πάνω από 10 ευρωπαϊκές χώρες έχουν υπάρξει απογραφές και ζητάμε να τεθεί τέλος στις φορολογικές διευκολύνσεις προς την, στην συγκεκριμένη δραστηριότητα. Επίσης από τις εξαιρέσεις για τα μέτρα για το περιβάλλον. Εμείς είμαστε υπέρ της δίκαιης φορολογίας, υπέρ της αρχής ότι αυτός ο οποίος μολύνει πρέπει και να πληρώνει. Ζητάμε επίσης την υπευθυνοποίηση των εταιριών αυτών απέναντι στο περιβάλλον, ε, και για την ευημε... τον σεβασμό του στην ευημερία των πολιτών σήμερα και στο μέλλον. Φαίνεται ότι οι αερομεταφορείς έχουν πετύχει μια κάποια ασυλία σε σχέση με τις αρχές αυτές. Τα αεροπορικά εισιτήρια δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ, τα καύσιμα των αεροσκαφών δεν πληρώνουν φόρο και δεν περιλαμβάνονται οι επιχειρήσεις στο σύστημα ε, εμπορίας καυσαερίων υπάρχουν κάποιοι φόροι αντικατάστασης του ΦΠΑ σε ορισμένες χώρες, αλλά είναι τόσο χαμηλή που δεν αξίζει να συζητάμε. Το αποτέλεσμα είναι πραγματικά απαράδεκτο. Κάποια βασικά προϊόντα όπως το ψωμί και το γάλα πληρώνουν πολύ περισσότερο φόρο από ότι οι ε, μεταφορικές εταιρείες, οι αεροπορικές εταιρείες. Και σύν της άλλης παίρνουν κρατική βοήθεια, κρατικές επιδοτήσεις, και πραγματικά αυτό αποδεικνύεται και από κάποιες τιμές εισιτηρίων οι οποίες είναι εκπληκτικά χαμηλές και προφανώς δεν καλύπτουν το στόχο. Υπάρχει ένα τεράστιο λόμπι μέσα από την ΙΑΤΑ και τα ΙΚΑΟ και το ΙΚΑΟ και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δημιουργεί στρεβλώσεις στον διεθνή ανταγωνισμό. Αν υποχρεώσει κανείς τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ε, με τις ε, υπόλοιπες εταιρείες, προφανώς ε, το φτηνό χρήμα των σεΐχιδων των αραβικών χωρών και το δωρεάν καύσιμο τους δίνει πλέον Θέλουμε όμως τέτοιου είδους καταστάσεις και για την Ευρώπη. Θα μπορείτε να μας πείτε μα τι γίνεται με τις θέσεις απασχόλησης, σαν παράδειγμα των αερομεταφορών. Η αλήθεια είναι ότι κάθε βιομηχανία θα μπορούσε να δημιουργήσει περισσότερες θέσεις απασχόλησης άμα δεν πλήρωνε καύσιμα. Και ο τρόπος με τον οποίο δημιουργούν θέσεις απασχόλησης ε, οι αερομεταφορείς ε, είναι λίγο περίεργος. Τους υπολογισμούς τους περιλαμβάνουν και τις δευτερευόντως σχετικές θέσεις απασχόλησης. Σαν παράδειγμα όταν ένας εργαζόμενος ας πούμε στην, σε μια επιχείρηση αγοράζει για την εταιρεία του κάποια έπιπλα τότε ο εργαζόμενος στην, στο κατάστημα των επίπλων θεωρείται ότι απασχολείται για την επιχείρηση. Αν όλες οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούσαν την ίδια μέθοδο τότε οι θέσεις που θα έπρεπε να υπάρχουν διαθέσιμες στην αγορά εργασίας θα ήταν περισσότερες από τους πραγματικούς εργαζομένους. Όπως λοιπόν λειτουργεί σήμερα η βιομηχανία η αεροπορική σαφώς και δεν συνεισφέρει στον προϋπολογισμό τον κοινοτικό, τον εθνικό και στους φοροϊσπρακτικούς μηχανισμούς. Αυτός είναι ο μηχανισμός ο οποίος κάνει τους πλούσιους πλουσιότερους και τους φτωχούς φτωχότερους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θέλει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Η οδηγία για το ΦΠΑ και η οδηγία για τον ενεργειακό φόρο ε, δίδουν πάρα πολλές εξαιρέσεις προς την βιομηχανία αυτή και η Επιτροπή δεν θέλει να το αλλάξει καθόλου. Το θέμα αυτό έχει παραπεμφθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα κράτη-μέλη, αλλά κανένα κράτος μέλος ε, μόνο του δεν θέλει να καταργήσει τα πλεονεκτήματα αυτής της βιομηχανίας και να θέσει να πάρει μέτρα όπως περιορισμού στις νυκτερινές πτήσεις και στον θόρυβο των αεροσκαφών. Είμαστε λοιπόν κατά κατηγορηματικά μιας αντιμετώπισης χώρα ανά χώρα γιατί δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Η Ευρωπαϊκή ε, Ένωση ρυθμίζει τις ε, βιομηχανίες, η γαστρονομία σαν παράδειγμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφασίζει αν το κάπνισμα επιτρέπεται στα, στα, ε, στα εστιατόρια και για το αν υπάρχουν αλλεργογόνα και αν πρέπει να αναφέρονται τα αλλεργογόνα στα τρόφιμα. Ε, για τον θόρυβο στα αεροσκάφη γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σφυρίζει αδιάφορα. Μήπως θα πρέπει εν πάση περιπτώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποφασίσει ότι οφείλει να δαμάσει τους ναι. αερομεταφορείς. Thank you very much for Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα θέλα τώρα να δώσω το λόγο στον Μάνφρετ Πράντε. Για τη δεύτερη <coughs> αναφορά για το θέμα αυτό. Χωρίς μικρόφωνο. Microphone, please. Oh, yes. Sorry. Συγγνώμη, εντάξει. Το όνομά μου είναι Μάνφρετ Πράντε, κατοικώ στην Κολονία. Είμαι παντρεμένος, συνταξιούχος 77 ετών και έχω δύο ενήλικα παιδιά. Επαγγελματικά ήμουνα μηχανολόγος ανάπτυξης σχεδιασμού αυτοκινήτων. Το καλοκαίρι 1969 και η οικογένειά μου και εγώ πήγαμε στη μονοκατοικία μας στο Κέρν Νόιμπερκ περίπου 7.300 μέτρα σε ευθεία γραμμή από τις, ε, τους διαδρόμους απογείωσης και προσγείωσης του αεροδρόμου Κέρν Βόνης, κολονίας Βόνης. Και ανάλογα με την κατεύθυνση του ανέμου ακολουθούν αυτούς τους διαδρόμους ε, τα ε, αεροπλάνα προσγειώνονται και μάλιστα σε ύψος 480-490 μέτρων ύψους ενώ οι, τα αεροπλάνα που ξεκινούν για να απογειωθούν δεν γνωρίζω σε ποιο ύψος κάνουν αυτό, ωστόσο δεν τηρούν ε, τις, ε, το εύρος των διαδρόμων τους και έτσι πολλές φορές παρεκκλίνουν και ο ήχος ή η χορύπανση ενοχλεί πολύ μεγαλύτερη, σε πολύ μεγαλύτερη ακτίνα. Παλιότερα μας ενοχλούσε η κίνηση στον αυτοκινητόδρομο, όμως με τυχώματα ε, αυτός ο θόρυβος μειώθηκε. Αντίθετα όμως αυξήθηκε ο θόρυβος από τα αεροπλάνα. Αυτό ισχύει κυρίως για μεγάλα εμπορικά αεροπλάνα που μεταφέρουν αγαθά που έχουν και πολύ υψηλό επίπεδο ηχητικής όχλησης 74 μέχρι 81 ε, ε, DBA και έτσι δεν μπορεί κανείς το βράδυ από τις 11 η ώρα έως τις 4.30 το πρωί να κοιμηθεί. Εδώ δεν πρόκειται μόνο για κάποιους ε, υπολογισμούς ηχητικής ρήπανσης, αλλά πραγματική ρήπανση. Η υγεία της γυναίκας μου και μου έχει υποστεί πλήγματα, δηλαδή έχουμε προβλήματα με την καρδιά μας, υψηλή πίεση, έχουμε TIA, δηλαδή περιοδικά επεισόδια ισχυμίας, παρότι δεν υπήρχαν τέτοια εικόνα ασθένειας οι γονείς μας. Προσπαθούμε να θεραπεύσουμε ή να καλύψουμε αυτές τις ανάγκες αυτών των ασθενειών εκτός κολονίας, ωστόσο πρέπει να αγοράζουμε και να καταναλώνουμε πολύ ακριβά φάρμακα. Το αεροδρόμιο κολονίας Βόνης βρίσκεται σε επεκτατική πορεία και θα υπάρχει όλο και μεγαλύτερη ηχητική ρήπανση, πράγμα το οποίο θα οδηγεί σε, αυξημένες, ε, ε, σε αυξημένα προβλήματα υγείας. Γραπτά και προφορικά παραπονεθήκαμε για αυτή την κατάσταση χωρίς όμως αποτέλεσμα. Επειδή οι αρχές, ε, οι των αεροδρομίων και οι πολιτικοί αναφέρονται πάντα σε κάποιους κανόνες και κανονισμούς που βρίσκονται πολύ μακριά από την πραγματική ζωή και δίνουν την ανώστατη προτεραιότητα στα οικονομικά συμφέροντα των αεροπορικών εταιριών. Δεν δίνουν καμιά σημασία στην προστασία των πολιτών εφόσον το αεροδρόμιο μπορεί να επιτύχει τους στόχους, τους στόχους του όσον αφορά θέσεις εργασίας και αυξημένα κέρδη με το τζίρο τους. Πραγματικότητα είναι ότι οι πολιτικοί και οι υπεύθυνοι των αεροδρομίων δεν ενδιαφέρονται καθόλου για να υπάρξει μια αντιστάθμιση συμφερόντων σε αυτήν την κατάσταση. Και βλέπουμε εδώ ότι τα όσα ε, πρόστιμα οι κυρώσεις ε, έχουν επιβληθεί δεν έχουν αλλάξει την κατάσταση. Οι εταιρείε μπορούν να πληρώνουν αυτά τα μικρά πρόστιμα και δεν επενδύουν έτσι σε λιγότερο ε, ε, ε, αεροπλάνα που προκαλούν ηχητική ρήπανση. Εγώ πιστεύω ότι η απαγόρευση συγκεκριμένων πτήσεων είναι αναγκαία προϋπόθεση για να προστατευτεί η υγεία των ατόμων εκείνων που πλήττονται από την ηχορύπανση. Ευχαριστώ. Thank you very much. Thank Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμβολή σας. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στους συναδέλφους, ε, τρεις, τρία ονόματα, κυρία Κουμπίτσα, η κυρία Πυρή και ο κύριος Ίχκα. Ποιος θέλει να πάρει το λόγο, εσείς θα το αποφασίσετε. Μίστερ Κουμπίτσα, εγώ είμαι ο κύριος Κουμπίτσα και θα ε, αναφερθώ με, στο θέμα της ε, φορολογίας και των ειδικών φόρων κατανάλωσης ε, και μετά οι συνάδελφοι θα συνεχίσουν με το θέμα του, με το τμήμα που αφορά το θόρυβο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε προσφάτως μία μελέτη τον Ιανουάριο του 2015 αναφερόμενοι συγκεκριμένα στο θέμα του ΦΠΑ, στο εναέριες μεταφορές και γνωρίζουμε ότι οι διεθνείς πτήσεις συγκεκριμένα δεν φορολογούνται σε κανένα από τα κράτη-μέλη, ενώ οι εσωτερικές πτήσεις ποτέ δεν απαλλάσσονται από φορολογία, εκτός από τέσσερα κράτη-μέλη. Επομένως το θέμα αφορά τις διεθνείς πτήσεις, όπου δεν υπάρχει ε, ΦΠΑ. Ε, υπάρχουν, ε, ε, υπάρχουν εξαιρέσει εξαιρέσεις που υπάρχουν από το 1977. Τα κράτη-μέλη έχουν τη δυνατότητα να συνεχίζουν τις εξαιρέσεις αυτές παρόλο που δεν είναι υποχρεωμένοι. Το 2016 όμως ανακοινώνουμε ένα καθεστώς 2016 και γι' αυτό ακριβώς αναφερόμαστε σε τέτοιου είδους απαλλαγές οι οποίες πλέον δεν θα είναι οριστικές στην απάντησή μα σας είχαμε δώσει τι σχετικέ αυτέ πληροφορίε. Υπάρχει και συνέχιση. Αυτή τη στιγμή έγινε ένα εργαστήριο φυσκάλη με τα κράτη-μέλη, με του κοινωνικού εταίρους και με τους εκπροσώπους του κλάδου. Αναφερθήκαμε συγκεκριμένα στο δικό σα επιχείρημα. Ειδικότερα για τη φορολογία των εισιτηρίων της αεροπορίας συζητήσαμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, σε σχέση με το γεγονό οτι ότι αλλάζει σιγά-σιγά η αγορά. Ε, θα υπάρξει υπάρξει τεράστια αύξηση των ε, μεταφορών των επιβατικών μέχρι το 2030 και βλέπουμε ότι αν υπάρχει ΦΠΑ σε ένα, με έναν κανονικό συντελεστή θα είχαμε 7,5% ε, μικρότερη εναέρια κυκλοφορία, ε, βέβαια εκπεφρασμένα σε επιβάτες ανά χιλιόμετρα. το 2010 είχαμε 217 3 εκατομμύρια επιβατών, ε, ε, επιβατικών χιλιόμετρων για θα πέσουμε σε 100, στα 175. Πρόκειται για ε, ένα από τα μέτρα, θα μπορούσαμε να μειώσουμε και κατά 4,5% τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα σε σχέση με το σενάριο κατά το οποίο δεν κάνουμε τίποτα. Πάντως η φορολόγηση ε, των, ε, πτήσεων, των διεθνών πτήσεων θα μπορούσε να γίνει, παρόλα αυτά δεν είναι το μοναδικό μέτρο που θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε. Α περάσουμε τώρα στη φορολογία των εισιτηρίων που υπάρχουν σε τουλάχιστον εξι κράτη-μέλη. Είναι δύσκολο να διαχωρίσει κανεί τη φορολογία από τις δαπάνες. Υπάρχουν πάντως έξι κράτη-μέλη που επιβάλλουν άμεσο φόρο στα εισιτήρια. Αποτελούν... Ε, συχνά μάλιστα ο φόρος ε, υπερβαίνει την τιμή του εισιτηρίου και υποθέτουμε ότι αντί των κανόνων που ισχύουν αυτή τη στιγμή για τις επιβατικές μεταφορές, όπου συμβαίνει αποτελεσματικά υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή, πτήση από τη Γερμανία στη Γαλλία, η Γερμανία και η Γαλλία μπορούν να φορολογήσουν, αλλά μόνο το κομμάτι που είναι πάνω από την επικράτειά τους. Ψάχνουμε λοιπόν για λύση που θα μπορούσε να δώσει στις ε, χώρες ε, ε, τη δυνατότητα φορολόγησης υπό των υφισταμένων κανόνων, όμως αυτά είναι τα ζητήματα που διακυβεύονται αυτή τη στιγμή. Θα το συζητήσουμε στην επόμενη ομάδα εργασία για το μέλλον του ΦΠΑ. Εκεί συζητούν τα κράτη-μέλη τι μελλοντικέ εξελίξει. Έτσι έχουν τα πράγματα. Έτσι επεξεργαζόμαστε το θέμα αυτό. Θα αρκεστώ σε αυτά που σας είπα και μετά τώρα θα περάσουμε ε, στον ειδικό φόρο κατανάλωσης που αφορά τα καύσιμα. Εγώ θα ήθελα να συνεχίσω με το θέμα της φορολόγησης. Ε, η φορολόγηση των καυσίμων ε, ε, καλύπτεται από την, από την Οδηγία 96 του 2003. Δεν υπάρχει πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αυτή τη στιγμή για τη φορολόγηση των καυσίμων. Παρόλα αυτά, σε δύο κράτη-μέλη όσον αφορά την εφαρμογή των υποχρεών απαλλαγών και δεδομένης της ομοφωνίας που χρειάζεται για τη φορολόγηση, έπρεπε να ληφθούν υπόψη αυτές οι δύο φωνές και η οδηγία που ισχύει αυτή τη στιγμή προβλέπει υποχρεωτική εξαίρεση για τη φορολόγηση των καυσίμων. Αυτά υπάρχουν στο εφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο. Πρώτο στοχείο, το κάθε κράτο μέλος μπορεί μόνο μερός να επιβάλλει ένα φόρο ε, για τις πτήσεις στα καύσιμα και για την ώρα μόνο ένα κράτη, κράτος μέλος, οι κάτω χώρες ε, το κάνουν σε γενικές γραμμές η Ιαπωνία και οι Ηνωμένε Πολιτείες. Δεν γνωρίζω άλλη χώρα να το κάνει. Παρ' όλα αυτά μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, μόνο ένα κράτος μέλος το κάνει. Δεύτερο θετικό σημείο του υπάρχοντος νομοθετικού πλαισίου είναι ότι όχι μόνο μονομερός αλλά και διμερός τα κράτη-μέλη μπορούν να συμφωνήσουν ε, επί τη βάση διμερού συμφωνίας να φορολογήσουν τις ενδοκινοτικές πτήσεις για την ώρα δεν υπάρχει ούτε μία τέτοια διμερή συμφωνία εντός της Ένωσης. Όσον αφορά τώρα την τρίτη ομάδα της διεθνής πτήσης ε, που, ως, που αναφέρονται ως προβληματικές, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεσμεύονται από διεθνείς συνθήκες όπως η Σύμβαση του Σικάγο και διάφορες άλλες διμερείς συμφωνίες ε, μεταξύ των ε, αεροπορικών εταιριών και των διεθνών οργανώσεων για την απαλλαγή από τη φορολόγηση χωρίς τα καύσιμα. Κάτι το οποίο λοιπόν σημαίνει ότι αν συμβεί οτιδήποτε εντό Ευρωπαϊκή Ένωσης μπορεί να φτάσουμε σε επίπεδο διεθνούς διατησίας και δεν μπορούμε να προβούμε σε αυτές τις αλλαγές. Μπορεί βέβαια η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταβάλει κάποιες προσπάθειες, είναι όμως μια μακροχρόνια διαδικασία και δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι στο άμεσο μέλλον θα ε, ολοκληρωθεί η προσπάθεια αυτή και θα καρποφορήσει. Εκτός από αυτά, ε, υπάρχουν, υπάρχει και κάτι ακόμη θετικό ε, το οποίο δεν έχει να κάνει τόσο με την νομοθεσία αλλά με τις αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ένωσης ε, που σε δύο αποφάσεις, τη Helmholtz και την Άντερ Μάουνσταφ έθεσε κάποιους, ορισμούς, ε, κάποιους περιορισμούς στην υποχρεωτική απαλλαγή ε, λέγοντας ε, ότι αφορά μόνο συγκεκριμένες υπηρεσίες. Όλα ε, τα αεροσκάφη που μεταφέρουν προσωπικό επιχειρήσεων δεν είναι υποχρεωμένες να προβαίνουν σε αυτή την απαλλαγή. Όπως σας είπα, το μόνο κράτος μέλος που, κάνει, που έχει, βάλει κάποιο είδους φορολογία είναι οι κάτω χώρες. Πρόταση για την αλλαγή της ε, φορολόγησης ενέργειας δεν ε, αποτελεί τμήμα του προγράμματος για, τον, ε, το επόμενο έτος και δεν ξέρουμε κατά πόσο θα γίνει και στο μέλλον. Είναι δύσκολο να κάνουμε μία πρόταση στο πλαίσιο ενός περιβάλλοντος όπου χρειάζεται ομοφωνία. Θα ήθελα τώρα να δώσω τώρα το λόγο στη συνάδελφο Ζουστίν Τιρέ. Έρχομαι από τη Γενική Εύθυνση Μουβ και καλύπτω το θέμα του θορύβου. Ο θόρυβος αεροπλάνα. Ο θόρυβος διαδραματίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στα αεροπλάνα. Και εδώ το γενικότερο πλαίσιο ε, είναι εκείνο το οποίο λειτουργεί και δεν μας δίνει τη δυνατότητα να προσαρμοστούμε σε ατομικές περιπτώσεις ξεχωριστά. Τα μέτρα που λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο είναι πάντα ευθύνη των κρατικών αρχών και όχι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εμείς προχωρούμε στην θέσπιση διαδικασιών και διεργασιών. Τώρα, όσον αφορά τις ε, εκπομπές ρήπων, μέσα στο πλαίσιο τώρα των εκπομπών, της εμπορίας εκπομπών ρήπων σε διεθνές επίπεδο η Ευρωπαϊκή Ένωση πάντα ήταν υπέρ του να υπάρχει ένα σφαιρικό πλαίσιο που να δίνει σφαιρική απάντηση για τις εκπομπές ρήπων. Εργάζεται σκληρά στην ICAO η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή στο, στην Διεθνή Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορίας ΔΟΠΑ, για να υπάρξει ένα πλαίσιο ορισμών και καθορισμών που θα δίνει τη δυνατότητα η ενιαία ρήπανση από αεροπλάνα να καλύπτεται. Τώρα θέλω να αναφερθώ στις νέες κατευθυντήρες γραμμές ε, όσον αφορά τους αερολιμένες ε, που τον Απρίλιο 2014 άρχισε να ισχύει ήταν ένα πολύ σημαντικό βήμα για τις αεροπορικές ε, μεταφορές ε, μια καλή ε, διασύνδεση όσον αφορά τα επίπεδα και της κινητικότητας των Ευρωπαίων πολιτών διασφαλίστηκε ενώ επίσης αποφεύγουμε τη στρέβλωση του ανταγωνισμού μέσα στο ενίο πλαίσιο με τους κανόνες που θεσπίζονται ένα ισοδίκαιο πλαίσιο θα ισχύει όσον αφορά τις ευρωπαϊκές εταιρείες εναέριων μεταφορών και τις ε, άλλες ε, αλλοδαπές εταιρείες εναέριων μεταφορών. Αυτά είχα να πω. Θα λάβει τώρα τον λόγο ο συνάδελφός μου από την Επιτροπή. Παρακαλώ. Καλό σας απόγευμα Μάρκο Παλιώτη είναι το όνομά μου. Θα ήθελα να μιλήσω για δύο λεπτά μόνο. Αλλά επειδή οι περισσότερες αναφορές που έχουμε ενώπιόν μας απόψε πρέπει να καλυφθούν, συμφωνήσαμε να υπάρχει η δυνατότητα, αν συμφωνείτε Πρόεδρε, να μιλήσω για κάποια λεπτά για να καλυφθούν οι πτυχές αυτές. Το μεγαλύτερο μέρος των απαντήσεων δηλαδή που ε, προσφέρουμε στις ε, περιπτώσεις αυτών των αναφορών. Πρώτα να αναφέρω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συνειδητοποιήσει απόλυτα τα προβλήματα και τη σπουδαιότητα της διασφάλισης της υγείας των πολιτών και των κινδύνων που εδώ ε, υφίστανται για την υγεία των πολιτών λόγω της συγχωρήπανσης ε, και ε, της ε, περιβαλλοντικής ρήπανσης. Υπάρχουν επιστημονικά τεκμήρια από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας που αφορά, αφορούν αυτά τα θέματα. Είμαστε σε επαφή με τον Παγκόσμιο Οργανισμό ε, Υγείας για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε καλύτερα αυτά τα νέα ευρήματα που δείχνουν ότι ίσως να υπάρχει κάτι περισσότερο εδώ από το αναμενόμενο. Τρία εκατομμύρια περίπου Ευρωπαίοι εκτίθενται σε κάποιο σημαντικό επίπεδο θορύβου. Αυτό δημιουργεί πρόβλημα, ενοχλεί τον ύπνο, επίσης τα παιδιά είναι δύσκολο να μπορέσουν να συγκεντρωθούν και να μελετήσουν και εκείνοι που έχουν καρδιαγγειακές ασθένειες υποφέρουν ιδιαίτερα. Υπάρχουν εκατοντάδες πρώιμοι θάνατοι στην Ευρώπη που συνδέονται με αυτό τους το ηχητικό επίπεδο της συγχωρήπανσης από τις αεροπορικές μεταφορές. Είναι ένα πρόβλημα που πολύ καλά γνωρίζουμε και το έχουμε συνειδητοποιήσει. Ευχαριστούμε τους συντάκτες των αναφορών, γνωρίζουμε όμως το, τη φύση του προβλήματος. Το ζήτημα είναι όταν ερχόμαστε στο ευρωπαϊκό επίπεδο νομοθεσίας και όχι στο εθνικό επίπεδο το νομοθετικό, δεν περιγράφονται επίπεδα η ούτε υποχρεώνονται τα κράτη-μέλη να τηρήσουν κάποιες διεργασίες. Αυτό είναι το στοιχείο κλειδί Αντίθετα, αφήνει την στάθμιση των διαφορετικών συμφερόντων στη διακριτική ευκαιρία των κρατών μελών, των κρατικών αρχών για συγκεκριμένη λήψη μέτρων ή δραστηριοποίηση κατά της, ε, των κινδύνων υγείας και ακριβώς λόγω των περιοίκων αεροδρομίων Αυτές οι αποφάσεις είναι απόλυτη αρμοδιότητα των κρατικών αρχών των κρατών μελών αναλαμβάνονται από αυτές. Έχουμε δύο οδηγίες την οδηγία πλαίσιο του 2449 για τις, ε, το επίπεδο ε, ηχορύπασης που αναφέρει ότι το κράτος μέλος ε, πρέπει να δράσει, να ταυτοποιήσει, να εντοπίσει την κατάσταση, να εντοπίσει τους κινδύνους στην υγεία αυτών των πολιτών και μετά πρέπει να υιοθετηθούν αναπενταετία προγράμματα δράσης τα οποία θα συζητηθούν και θα αναλυθούν και έτσι ο πληθυσμός, οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να παρέμβουν με τις παρεμβάσεις τους. Και αυτό κύριο κέριο σημείο. Και πάλι όμως η τελική απόφαση είναι των αρμόδιων εθνικών κρατικών αρχών και όχι των ευρωπαϊκών αρχών ακόμα και στις αναθεωρήσεις, ε, επανεξετάσεις, οι εθνικές αρχές των κρατών μελών θα αποφασίζουν ποια συγκεκριμένα μέτρα θα πρέπει να λαμβάνονται. Τώρα, για την υπέρβαση εθνικών τέτοιων ε, ορίων και για την ευθυγράμμιση με, ε, ευρωπαϊκά, με ευρωπαϊκές τέτοιες τιμές, αυτό αφορά αποφάσεις και μηχανισμούς εθνικού επίπεδου που εκεί χρησιμοποιούνται τα στοιχεία για την ε, θέσπιση ενός κρατικού προγράμματος ε, δράσης. Να δούμε ποια μέτρα δηλαδή ή σύνολο μέτρων απαιτούνται. Πάλι εθνική αρμοδιότητα των κρατών μελών, των αρχών των κρατών μελών. Συμπεραίνουμε και πάλι ότι οι παράγοντες αυτοί που αναφέρονται στις αναφορές ε, επανειλημμένα απαιτούν οι πολίτες να ενημερώνονται σωστά με, σε σχέση με τη μεθοδολογία υπολογισμού συντελεστών κινδύνων όμως ε, επαφίεται στις, αρχι... στις κρατικές αρχές των κρατών μελών να αποφασίσουν το τι θα ισχύει και για το τι θα ισχύσει και για τον αντίστοιχο κανονισμό 598 ε, ναι, του 2014 που θεωρήθηκε ότι θα είναι ο μηχανισμός που θα αποφεύγει να υπάρχουν θα, για την απαγόρευση δηλαδή πτήσεων ή χορύπασης δεν συμβαίνει όμως αυτό δημιουργείται μόνο μια δομή από αυτόν τον κανονισμό για τις αποφάσεις που θα λαμβάνονται και τη διαδικασία που θα ακολουθείτε και το επαναλαμβάνω για τελευταία φορά η τελική απόφαση, η καθοριστική απόφαση εξακολουθεί να βρίσκεται και είναι αρμοδιότητα των εθνικών κρατικών αρχών των κρατών μελών. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για την ε, παρουσίαση αυτών των θεμάτων τα οποία θα μας απασχολήσουν απόψε. Ευχαριστώ. Αρχίζει τώρα ο γύρος παρεμβάσεων των συναδέφων. Ποιοι θέλουν να παρέμουν παρακαλώ για αυτό το θέμα. Εσείς κύριε έχετε τον λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Υπάρχουν ε, συμφέροντα από δύο πλευρές στη συγκεκριμένη περίπτωση. Από τη μία μπορεί να το δει κανεί σαν την επιθυμία των αερομεταφορών να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους και από την άλλη υπάρχουν ε, αυτοί οι οποίοι πιστεύουν ότι θα πρέπει τα κακώς κατά αυτούς κείμενα να διορθωθούν. Οι διεθνείς κανονισμοί μπορεί να ρυθμίζουν τα θέματα της ασφάλειας στις αερομεταφορές. Και από την άλλη πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν ε, σε σχέση με τις χωροτακτικές ρυθμίσεις οι οποίες γίνονται γύρω από τους αερολιμένες ε, αρμοδιότητες οι οποίες είναι καθαρά εθνικές και οι εθνικές υπηρεσίες είναι αυτές οι οποίες θα προσπαθήσουν να υπολογίσουν αξιολογώντας ε, ένα αίτημα ε, ποιο θα είναι το ποσό το ανεκτό της μόλυνσης είτε ηχητικής είτε χημικής. Δεν βλέπω λοιπόν πώς μπορούμε εμείς να παρέμβουμε. Αυτή είναι μια αναφορά η οποία θα πρέπει να αποσταλεί στα εθνικά κοινοβούλια οι οποίοι θα πρέπει να ελέγξουν αν υπάρχουν λάθη στους νόμους που άπτονται της χωροταξίας των αερολιμένων. Έτσι λοιπόν θα πρέπει οι επενδύσεις στον τομέα αυτό να αξιολογούνται έτσι ώστε να ελέγχεται αν δημιουργούνται προβλήματα στους γείτονε των αεροδρομίων οι οποίοι μπορεί να υποφέρουν. Εγώ δεν γνωρίζω τις ε, εθνικές ε, αν θέλετε ρυθμίσεις. Εγώ γνωρίζω τι συμβαίνει στην Πολωνία, τι κάνει η κυβέρνηση αν υπάρξει ένα θέμα. Έχουμε και εμείς ένα πρόβλημα στην Πολωνία με ένα αεροδρόμιο το οποίο βρίσκεται κοντά σε πόλη ε, το κράτος είναι αυτό το οποίο είναι αρμόδιο, το οποίο θα ελέγξει εάν πράγματι ε, χρειάζεται να μετακινηθούν κάποιοι άνθρωποι σε διαφορετικές περιοχές και το κράτος έπαιξε το ρόλο του και τώρα το πρόβλημα στη χώρα μου έχει αντιμετωπιστεί. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω ίσως ε, ε, οι αναφερόμενοι αν έχουν προβεί σε διαβήματα στο εσωτερικό των χωρών τους. Επαναλαμβάνω, πιστεύω ότι είναι εθνικό θέμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν θα ήθελε κάποιος άλλος το λόγο. Εύη. Ευχαριστώ πολύ. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα αυτό και ευχαριστώ όλους τους αναφερομένους που το έθεσαν με τόσο εύγλωπο τρόπο. Θα ήθελα να εκφράσω εδώ μια γενική ε, σκέψη. Θα ήθελα να αναφερθώ ειδικότερα όμως πρώτα στο θέμα του ETS. Το σύστημα των αερομεταφορών δεν καλύπτεται πάντα από το σύστημα εμπορίας εκπομπών καυσαερίων και όμως είναι ένας τομέας στον οποίο είναι προφανές ότι το σύστημα ETS αφ' αυτού έχει αποτύχει. Ξέρετε ότι η τιμή των μερισμάτων του συστήματος αυτού είναι στην ελεύθερη αγορά ε, πραγματικά πάρα πολύ χαμηλά και δεν θα φτάσει τα 35-36 ευρώ αναμέρισμα που θα ήταν απαραίτητο για να χρηματοδοτηθεί η πορεία προς τεχνολογίες πολύ πιο αηφόρες και σε σχέση με το περιβάλλον. Λοιπόν, αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι επίσης η επιρροή ε, του ETS ε, στο εισιτήριο είναι κάτι το οποίο αναλαμβάνει πλήρως ο καταναλωτής και δεν λαμβάνεται υπόψη ε, η βασική αρχή η οποία λέει ότι αυτός ο οποίος μολύνει είναι αυτός ο οποίος θα πρέπει να πληρώνει το κόστος το οποίο προκαλείται. Ελπίζω να υπάρξουν κάποιες βελτιώσεις από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής γιατί έχουμε μπροστά μας ένα πρόβλημα θεμελιώδες το οποίο αφορά όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί να μην εφαρμόζεται εδώ οι, οι βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι δεν πληρώνουν ουσιαστικά τίποτα από το κόστος που τους αναλογεί για τη μόλυνση οι αεροπορικές επιχειρήσεις με τον τρόπο αυτό δεν προστατεύεται όπως θα έπρεπε να προστατεύεται η ανθρώπινη υγεία και φυσικά το περιβάλλον. Γιάρεκ, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συμφωνώ με τους αναφερομένους. Εμείς εδώ στην Επιτροπή μας πρέπει να δώσουμε μία απάντηση ουσιαστική έχει υπάρξει παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας. Από ό,τι λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει υπάρξει κάτι τέτοιο. Ως εκ τούτου είναι πάρα πολύ δύσκολο για μας να δώσουμε συνέχεια σε αυτές τις αναφορές. Καταλαβαίνω τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι συγκεκριμένοι κάτοικοι των περιοχών γύρω από τα αεροδρόμια, αλλά διαρωτώ με εμείς τι μπορούμε να κάνουμε γύρω από αυτό. Okay, I don't have anybody else. Δεν βλέπω κανέναν άλλο να θέλει να πάρει το λόγο. Ωραία, αυτό που θα μπορούσαμε να κάνουμε είναι το εξή. Κανένα δεν πρότεινε τίποτα. Οπότε κάπως πρέπει να συνοψίσω. Γιάρεκ, θες να προτείνεις κάτι. Λοιπόν, προτείνω να κλείσουμε αυτές τις αναφορές. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Δεν υπάρχει παραβίαση της ε, ενωσιακής νομοθεσίας. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Επιτέλους κάποιος πρότεινε κάτι συγκεκριμένο. Αυτό χρειάζομαι. Δεν ε, μπορώ να βγάλω συμπέρασμα χωρίς τη συμβολή των συναδέλφων. Λοιπόν, προτείνω το εξής. Για να μετριάσω κάπως τη σκληρότητά σας. Εγώ λέω να, να στείλουμε στις επιτροπές ΕΜΒΙ και ΤΡΑΝ ε, το θέμα προς ενημέρωσή τους και να ζητήσουμε ενδεχομένως και μία γνωμοδότησή τους. Ίσως θα ήταν καλύτερα να αποστείλουμε μια ενημερωτική επιστολή στις επιτροπές αυτές ότι είναι ένα ζήτημα που ανησυχεί πολλούς πολίτες, ότι δεν παραβιάζει τις ε, οδηγίες της Ένωσης. Είναι ένα θέμα το οποίο ε, διέπεται από την επικουρικότητα και ε, εθνική αρμοδιότητα. Παρόλα αυτά αποτελεί τεράστια ανησυχία για πολλούς Ευρωπαίους πολίτες. Οπότε πιστεύω ότι οι Επιτροπές Περιβάλλοντος και Μεταφορών θα έπρεπε να γνωρίζουν ότι υπάρχει αυτή η πρωτοβουλία ε, ε, του ελέγχου της αεροπορίας, ε, ότι είναι κάτι που έχει προσελκύσει την προσοχή πολλών πολιτών, πολλών συμπολιτών μας και εμείς από την πλευρά μας μπορούμε να κλείσουμε την αναφορά αυτή και να το προωθήσουμε στις νομοθετικές επιτροπές. Συμφωνείτε? Πολύ ωραία. Λοιπόν, τότε συνεχίζουμε με, το, με τις πτήσεις και περνάμε στην αναφορά 0274-2012 των Φόλκερ Χάμπλ και Rudolf Μπραντ συνοδεύεται από περίπου 320 υπογραφές για την ηχορύπανση από τις νυχτερινές πτήσεις ε, που εκτελούνται στον αερολιμένα της ε, Φραγκφούρτης στη Γερμανία. Δεν είναι εδώ οι αναφέροντες, αλλά είναι εδώ εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οπότε θα τους δώσω το λόγο. Yeah. Thank you. Uh, Ευχαριστώ. Θα ήθελα να αναφερθώ και στα... να σας παραπέμψω στα προηγούμενα μας σχόλια. Yeah. Για την προηγούμενη αναφορά δεν έχουμε τίποτε να προσθέσουμε. The floor is open to colleagues. Συνάδελφοι, θέλει κανείς το λόγο? Ωραία. Υποθέτω ότι θέλετε να κάνουμε το ίδιο και για την προηγου... που κάναμε και την προηγούμενη αναφορά. Να αποστείλουμε στις επιστολές Τραν και Έμβη ε, ενημερωτική επιστολή για να την κλείσουμε την αναφορά. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε να προσθέσω ότι σχετικά με την Επιτροπή Περιβάλλοντος και μετά από αυτά τα οποία μας είπαν οι συνάδελφοι και η Επιτροπή εδώ, έχουμε να κάνουμε με θέματα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά όχι μόνο για τους ίδιους τους πολίτες αλλά και για μας τους νομοθέτες. Έχουμε να κάνουμε δηλαδή με μια νομική ρύθμιση ήδη από το 2014 όπου τέθηκαν τα θέματα αυτά. Σχετικά αναφέραμε ειδικότερα στο θέμα της ηχητικής, της ηχητικής μόλυνσης. Όπως είπε και η συνάδελφος κυρία Εύη, περιμένουμε την αναθεωρημένη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εγώ παρακολουθώ προσωπικά τις συναντήσεις ε, για το κλίμα που είχαν ξεκινήσει στην Κόπενχάγη σε συνεργασία με τον κύριο Λίζε έχουμε συναντηθεί επανειλημμένα με εκπροσώπους της ΙΚΑΟ και μπορώ να σας μεταφέρω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει προσπαθήσει να μεταφέρει προς το ΙΚΑΟ τον καπτεπίγοντα χαρακτήρα του αιτήματο αυτού των πολιτών. Πρόκειται για ένα σύστημα το οποίο είναι ιδιαίτερος παγκοσμιοποιημένο και γι' αυτό ακριβώς απαιτείται σε παγκόσμιο επίπεδο να υπάρξουν ε, οι απαιτούμενες ρυθμίσεις. Ε, κάποια πρώτα βήματα έχουν γίνει, ίσως να μην είναι τόσο αν θέλετε συγκεκριμένα όσο θα περίμενε κανείς, αλλά είναι σαφές ότι το ΙΚΑΟ έχει αρχίσει να συνειδητοποιεί την σημασία που έχει το θέμα. Είναι σωστό να παραπέμψουμε το θέμα αυτό στην, ε, ε, στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή, αλλά είναι τυπικό σαν βήμα, δεν είναι ουσιαστικό, δεν αναφέρεται στις αρμοδιότητες μας, στις κατεξοχήν, ε, θα έλεγα, σημαντικές που έχουμε στον συγκεκριμένο τομέα. δεν ξέρω αν μπορούμε να κρυφτούμε πίσω από το ότι πρόκειται για αποκλειστική, όπως λέγεται, εθνική αρμοδιότητα. Αυτό που είναι σαφές είναι ότι με μεγάλη αυτή τη στιγμή προσπάθεια και η προσπάθεια αυτή δεν θα πρέπει να περιορίζεται σε αυτό το οποίο είπατε. Ότι δηλαδή να παραπέμψουμε τις αναφορές όλες αυτές στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές. Δεν είμαι αντίθετη με αυτό, αλλά δεν φτάνει αυτό μόνο. Είναι κάτι το τυπικό. Κατά πάσα πιθανότητα ναι. Έτσι μπορούμε να δείξουμε στις νομοθετικές επιτροπές ότι είναι κάτι που προκαλεί μεγάλη ανησυχία σε πολλούς Ευρωπαίους πολίτες. Γι' αυτό δεν είναι αρκετό να γίνει απλώς η ακρόαση εδώ και ε, να ακούσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας λέει μια φορά ότι δεν παραβιάζεται Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Αυτό μπορούμε να κάνουμε και μπορούμε βεβαίως ε, ως ομάδες, ως μεμονωμένοι ε, ευρωβουλευτές να το προωθήσουμε το θέμα σε σεμινάρια, ημερίδες ή οτιδήποτε, αλλά ε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε άλλο στην Επιτροπή μας. Λοιπόν, θα στείλουμε ενημερωτική επιστολή στις Επιτροπές Μεταφορών και Περιβάλλοντος και θα κλείσουμε την αναφορά αυτή. περνάμε τώρα στο 14, επειδή πρόκειται για γαλλικό ε, σε, για γαλλικό ε, θέμα και μετά θα επιστρέψουμε στο 13. Είναι εδώ οι αναφέροντες. Καλώς ήρθατε. Εμμανουέλ Λετεξιέ και Αντουάν Λεμί. Και σας δίνω το λόγο. Ευχαριστώ, Αντουάν Φιλελμή και είμαι μέλος ε, της ε, οργάνωσης Πακεστιόν, Επουδενή, και θα σας μιλήσουμε για τις ε, Βρυξέλλες. Εμείς έχουμε να αντιμετωπίσουμε μία μοναδική κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μία πολιτική κατακαιρματισμού και ε, Παράκαμψη ε, των πολιτών αεροσκαφών πάνω από τι πιο πυκνοκατοικημένε περιοχές. Πάνω από ένα εκατομμύριο άτομα πλήττονται. Οι Βρυξέλλε, ε, από απόψε ως συγκριτικής αξιολόγησης είναι ο χειρότερος μαθητής όσον αφορά τη διαχείριση της συγχωρήπανση και μιλάω για τις Βρυξέλλες. Η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί για να μεγιστοποιεί τους ανθρώπους που πλήττονται από τις υπερπτήσεις και δεν υπάρχει αποζημίωση. Νυχτερινές πτήσεις περνούν από το 1988 ε, πάνω από τουλάχιστον 480.000 άτομα στο κέντρο των Βρυξελών. Υπάρχουν εναλλακτικέ επιλογές, υπάρχουν προγράμματα τα οποία επιτρέπουν να μειωθεί ο αριθμός των θυμάτων ηχορύπανση κατά πάνω από 72% και εδώ στο κέντρο ε, των ε, θεσμικών οργάνων της Ένωσης τίποτε δεν γίνεται από το κράτος του Βελγίου υπάρχουν παραβιάσεις, ε, υπάρχει τεράστια παραβίωση της οδηγίας 49 ε, του 2002 και θα σας αφήσω την κυρία Τεξιέ να σας εξηγήσει. Ναι, από τις 6 Φεβρουαρίου 2014 ε, το πρόγραμμα ε, παράκαμψη των πτήσεων ήταν, ε, προκάλεσε τεράστια ανησυχία στους ε, πολίτες και έφτασε μέχρι τα βελγικά δικαστήρια και θα ήθελα να πω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι προφανώς δεν γνωρίζετε τις τελευταίες εξελίξεις γιατί υπάρχει μια διαταγή από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο στις 31 Ιουλίου του 2014 που διέταξε τη διακοπή των δρομολογίων που άρχισαν το Φεβρουάριο του 2014. Το Βέλγιο μόνο εν μέρη έχει εκτελέσει αυτό το διάταγμα και έκανε μάλιστα και προσφυγή. Η χορύπανση από το αεροδρόμιο των, Βρυξεκόλ, ε, των Βρυξελών δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα ε, στους πολίτες και ε, παραβιάζει την ενωσιακή νομοθεσία. Βλέπετε πόσο μεγάλη είναι η παραβίαση για μας ε, η οδηγία 49 ε, του 2002 παραβιάζεται συνεχώς από το ε, Βέλγιο. Σας υπενθυμίζω ότι αυτή η οδηγία προ προβλέπει ότι πρέπει να υπάρξει σχέδιο δράση για τη μείωση του θορύβου στις περιοχές γύρω από τα μεγάλα αεροδρόμια. Άρθρο 8 παράγραφος 5 η οδηγία αναφέρει ότι επαφίεται βέβαια στις αρμόδιες αρχές πώς θα συμβεί αυτό αλλά θα έπρεπε να υπάρχουν προτεραιότητες για να μην γίνεται και υπέρβαση των σχετικών οριακών τιμών. Αυτή η οδηγία κατά κάποιο τρόπο μετεγράφει στη βελγική νομοθεσία, όμως αναποτελεσματικά οι Βρυξέλλες, η Βαλονία και η Φλάνδρα έχουν ε, περιβαλλοντική αρμοδιότητα, ενέκριναν μια νομοθεσία επιτόπου, με... άρχισαν κάποια προγράμματα διαχείρισης, αλλά το Βέλγιο έχει την αρμοδιότητα διαχείρισης εναέρης κυκλοφορίας και καθορίζει τα δρομολόγια και δεν επιτρέπει στις περιφέρειες να προβούν στα σχέδια και ε, στέλνει τα αεροπλάνα πάνω από την περιφέρεια των Βρυξελών, ε, κάτι το οποίο σημαίνει τεράστια επίπεδα θορύβου. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ε, από τις 6 μέχρι τις 7 το πρωί έχουμε τεράστιες υπερβάσεις ε, των σχετικών ορίων. 45 ε, ε, δεσιμπέλ είναι το, το, το όριο και 9 στα 10 ε, μηχανήματα μέτρησης του θορύβου περνάνε τα 65 δεσιμπέλ κατά τη διάρκεια της ε, περίοδου αυτής, 6 με 7 το πρωί. Ε, στις 23 ε, Ιουλίου ε, ζητήθηκε ενημέρωση του προγράμματος διαχείρισης του θορύβου όπως πρέπει να γίνεται κάθε πέντε χρόνια και πρέπει να υπάρξει διαβούλευση με τον πληθυσμό. Ζητούμε και άλλα μέτρα που πρέπει να ζητηθούν από την Επιτροπή Αναφορών να μην κλείσει αυτή η αναφορά. Αυτή τη στιγμή η ενημέρωση αυτών των τριών περιφερειών του Βελγίου δεν έχει ολοκληρωθεί και αυτή τη στιγμή δεν έχει ολοκληρωθεί και η υπόθεση στο δικαστήριο να υπάρξει μια έρευνα για τους λόγους για τους οποίους το Βέλγιο δεν εφαρμόζει το πρόγραμμα διαχείρισης που επιτάσσει η οδηγία από το 2002 και παρεμποδίζει την περιφέρεια των Βρυξελών από ε, την εφαρμογή του προγράμματος αυτού. Θα θέλαμε λοιπόν να ζητήσουμε το σεβασμό ε, από το Βέλγιο της οδηγίας 2002. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ και δίνω το λόγο απευθείας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Yes, thank you. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Όσον αφορά το πρόγραμμα δράσης για τις Βρυξέλλες, βρίσκεται στο δημόσιο τομέα το θέμα και ζήτησε η Επιτροπή από τις αρμόδιες ευελικέ ε, αρχέ, γιατί δεν υπάρχει πρόγραμμα δράσης, πώς στοχεύουν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα, τι θα ισχύει στις Βρυξέλλες και στο Βέλγιο όσον αφορά περιφέρειες και ζήτησε διευκρινήσει γενικά. Πρόεδρος. Πρέπει να πω ότι είναι κάπως αστείο ότι όταν είπατε ότι σε τρεις περιφέρειες ίσως κατά κάποιο τρόπο ε, ορίζονται αυτά. Η, ε, το Βέλγιο δεν είναι ένα απροσκεντροποιημένο κράτος. Είναι όμως ενδιαφέρον αυτό το οποίο μας λέτε. Ανοίγει τώρα ο διάλογος μεταξύ ευρωβουλευτών. Πρώτα απ' όλα έχουμε την Ελεονόρα Εύη, παρακαλώ, και μετά ο Γιάρεκ ε. Να μου επιτρέψετε να αναφερθώ και σε αυτήν και στην προηγούμενη αναφορά. Δεν νομίζω ότι το κλείσιμο των αναφορών αυτών είναι κάτι το κατάλληλο. Τι εννοώ. Είναι σαφές ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα ευρωπαϊκά όργανα αναζητούν να προσπαθήσουν περιπτώσει να βελτιώσουν την εφαρμογή των οδηγιών και σχετικά με τις μεταφορές και σχετικά με τις κλιματολογικές αλλαγές. Αλλά χάρη ακριβώς σε αυτές τις καταγγελίες αναφορές των πολιτών έχουμε για μια ακόμη φορά θα έλεγα την υποχρέωση να δούμε ακριβώς την παρούσα φάση το τι ισχύει γύρω από το θέμα της εφαρμογής των οδηγιών. Είναι αληθές ότι επικρατούν καταστάσεις οι οποίες είναι ε, εθνικής αρμοδιότητας όπου ασκεί η αρχή της επικουρικότητας και τα κράτη-μέλη, τα μεμονωμένα κράτη-μέλη είναι αυτά τα οποία θα πρέπει να προχωρήσουν στην εφαρμογή ε, των διατάξεων για τη μείωση του θορύβου στα αεροδρόμια. Είναι επίσης αληθές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει ε, εν πάση περιπτώσει να λειτουργήσει ελεγκτικά σε σχέση με τις ακολουθούμενες ε, διαδικασίες. Γιατί αν οι πληθυσμοί ε, οφείλεται να ενημερώνονται, και αυτό είναι κάτι το, για το οποίο εμείς επιμένουμε, είναι κάτι το οποίο υπογραμμίζουμε έντονα, θέλουμε να υπάρχει μια δημόσια εμπλοκή σε σχέση με τα θέματα αυτά Γι' αυτό λοιπόν και εγώ θα περίμενα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει ένα περιθώριο δράσης και να μπορέσει να πιέσει εν πάση περιπτώσει τα κράτη-μέλη να λειτουργήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Γιατί έχω την αίσθηση ότι πίσω από το άλοθη της επικουρικότητας εγκαταλείπουμε τους πολίτες οι οποίοι δεν ε, κάνουν τίποτα άλλο από το να βλέπουν ότι τα ευρωπαϊκά όργανα είναι ιδιαίτερος μακριά τους και δεν ασχολούνται καθημερινά με τα προβλήματα τα οποία αυτοί αντίθετα ζουν σε καθημερινή βάση. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξουν κάποιες ε, εθνικές ρυθμίσεις, αλλά αν οι ρυθμίσεις αυτές ε, δεν υπάρχουν, δεν είναι δυνατόν να λέμε ότι δεν υπάρχει τίποτα το οποίο μπορούμε να κάνουμε. Κοιτάξτε, αυτή είναι διαφορετική αναφορά. Ε, εντάσσεται πλέον στο θέμα της ευρωπαϊκής αρμοδιότητας, γιατί υπάρχει από πέρυσι ένας νέος κανονισμός, το 558 του 14, για τον καθορισμό κανόνων και διαδικασιών σχετικά με την εισαγωγή περιορισμών σχετικών με την ηχομόλυνση στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια. Ανακαλείται η προηγούμενη οδηγία. Ε, στο άρθρο 8 συγκεκριμένα αυτής της νέας οδηγίας υπάρχει υποχρέωση δημιουργίας καταρχάς ε, οργάνωσης μιας δημόσιας διαβούλευσης ιδιαίτερα για το αεροδρόμιο του Ζάβεντε που ξεκίνησε ήδη από το 2010. Μιλάμε για μια διαφορετική αναφορά και θα πρέπει τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν την διαδικασία που προβλέπεται τώρα. Αυτά τα οποία είπαμε πριν ισχύουν για τις άλλες αναφορές, όχι όμως για αυτήν. Αυτή ακριβώς ήταν και η πρόθεσή μου να υπογραμμίσω το ότι εμείς οφείλουμε να υπογραμμίσουμε την δημόσια διαβούλευση και την συμμετοχή του κοινού στον καθορισμό αυτών των προγραμμάτων. Είναι σαφές ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, θα πρέπει να μας δώσει μια ξεκάθαρη σε σχέση με αυτό απάντηση. Η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν ήταν επαρκής. Θα πρέπει λοιπόν να μας ενημερώσει καλύτερα για το πώς ασχολούνται οι βελγικές αρχές με την καινούργια οδηγία και ιδιαίτερα με το άρθρο 8 της νέας οδηγίας, το οποίο λέγει ότι η διαβούλευση με το κοινό θα πρέπει να ολοκληρωθεί. Εμείς δεν έχουμε πάρει καμία απάντηση σε σχέση με αυτό. Απαιτείται λοιπόν να το κάνουμε. Γιάρεκ, θες να πεις κάτι? να αναδιατυπώσω αυτό που είπες. Έχουμε τον κανονισμό 597 ε, βάση του οποίου ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο το οποίο πρέπει να επιβάλλει να εφαρμόζεται στα κράτη-μέλη. Τώρα όμως ο Βέλγος, ε, οι βελγικές αρχές πρέπει να τοποθετηθούν. Τι πρέπει να κάνουμε, αν υπάρχει ενωσιακή νομοθεσία που πρέπει να εφαρμοστεί, πρέπει να ζητήσουμε να γίνει αξιολόγηση από το βελγικό κράτος κατά πόσο εφαρμόζεται όντως αυτή η διαδικασία της διαφούλευσης με ε, τους πολίτες από τις βελγικές αρχές. Για να μπορέσει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας δώσει καλύτερες πληροφορίες για την επόμενη φορά, γραπτός ενδεχομένως, ε, θα έχουμε και συνεχή διάλογο μαζί σας και εμείς ως Επιτροπή θα... Ε, γράψουμε στις βελγικές ε, αρχές και θα του ζητήσουμε περισσότερες πληροφορίες για την αξιολόγηση θορύβου που πρέπει να, γίνουν, να γίνει στο πλαίσιο αυτής της διαβούλευσης για το σχέδιο δράσης του αεροδρομίου του Ζάβεντεμ ε, ε, η οποία αποφασίστηκε το 2010 και κατόπιν απόφαση του δικαστηρίου. Και θα το στείλουμε βέβαια ενημερωτικά και στις Επιτροπές Μεταφορών και Περιβάλλοντος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να πάρει το λόγο. Ναι. Εμείς θα προτιμούσαμε σε ένα λεπτό να διευκρινίσουμε λίγο περισσότερο τα πράγματα γιατί απλώς ε, μετά θα κάνουμε μια ανταλλαγή πληροφοριών γραπτών και δεν θα υπάρχει σαφήνεια. Ε, δεν θέλω να σας προσβάλλω, αλλά υπάρχουν ε, τρεις νόμοι. Η 49 του 2002 που λέει ότι οι πολίτες πρέπει να συμμετέχουν στη συζήτηση κάθε φορά που ένα σχέδιο δράσης ε, αποφασίζεται. Αυτό το σχέδιο δράσης πρέπει να αναθεωρείται κάθε πέντε χρόνια. Κάθε πέντε χρόνια λοιπόν θα πρέπει να γίνεται αναθεώρηση. Όσον αφορά τα μέτρα και συγκεκριμένα την απαγόρευση των πτήσεων είτε πρόκειται για τα πιο θορυβόρια αεροσκάφη ή για το κλείσιμο των ε, νυκτερινών πλήσεων, την απαγόρευσή τους, υπάρχει η, οδηγία 30 του 2002 και ο κανονισμός του 598 του περσινού έτους που θα αρχίσει να ισχύει το 2016. Όσον αφορά λοιπόν τη διαδικασία για, του περιορισμού ή την απαγόρευση των πτήσεων, μόνο λοιπόν για τον περιορισμό των πτήσεων και για κανένα άλλο μέτρο, τότε πρέπει να ακολουθείτε μία νέα διαδικασία. Δεν είναι απλώς ότι μία αρμόδια αρχή αποφασίζει, αλλά πριν λάβει την απόφαση πρέπει να γίνει μία διαβούλευση και πρέπει να γίνει μία αξιολόγηση των οικονομικών συνεπειών κλπ βάσει μιας ε, γνωμοδότησης από μια ανεξάρτητη αρχή. Σας το λέω αυτό απλώς διευκρινητικά γιατί λαμβάνουμε τα σχόλια από τους αναφέροντες και πρέπει να προσπαθήσουμε να διευκρινίσουμε για να μην χρειάζεται να κάνουμε ανταλλαγή απόψεων άχρηστη. Προφανώς και διευκρινίσατε σε μεγάλο βαθμό παρόλα αυτά πρέπει να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά. Αυτό είναι το πρώτο και πρέπει να δούμε τι θα γίνει. Πιστεύω ότι πρέπει να αποστείλουμε μια επιστολή στις βρυγικές αρχές για να τις ρωτήσουμε πώς προτίθενται να συνεχίσουν με τη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης και να ε, γίνει βέβαια και η επιστολή στις άλλες επιτροπές όπως ανέφερα για να γνωρίζουν ότι αυτό έχει προσελκύσει τεράστια προσοχή ε, από τους ε, Ευρωπαίους ε, πολίτες και δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε. Θα υπάρξει βέβαια και συνέχεια, θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό. Τώρα, πάμε στην αναφορά του κυρίου Λαβριέ ε, 1484 του 2008 είναι μια παλιά αναφορά όσον αφορά τις επιπτώσεις ηχητικής και ατμοσφαιρικής ρήπανσης στην υγεία των κατοίκων που διαμένουν πλησίων του αεροδρομίου Charles de Gaulle Roissy. Είναι εδώ η αναφέρουσα. Κυρία Κατρίν Λεκόντ. Σας δίνω το λόγο. Για μια στιγμή παρακαλώ. Η κυρία Εύη έχει ζητήσει πρώτα το λόγο. Ένα δευτερόλεπτο μόνο κανονικά. Δίνουμε ξανά το λόγο στους αναφερομένους μετά από την παρουσίασή τους. Ίσως για αυτούς των οποίων η αναφορά έκλεισε. Κανονικά θα έπρεπε να τους δώσουμε το λόγο για να απαντήσουν πριν περάσουμε στο επόμενο θέμα. Έχετε απολύτως δίκιο. Σκεφτήκα ότι μιας και όλοι οι αναφερόμενοι είναι στην αίθουσα, σκέφτηκα να ακούσουμε κάποιες αναφορές και μετά να πάρουν την δυνατότητα να το σχολιάσουν γιατί πιστεύω ότι τα θέματα αυτά είναι ιδιαίτερη σημασία όχι μόνο για τους παρόντες αναφερομένους αλλά και για το σύνολο του πληθυσμού. Έπρεπε να σας ζητήσω από την αρχή να ξαναπάρετε το λόγο. Ας ακούσουμε λοιπόν τώρα την επόμενη αναφορά. Έχετε το λόγο, κυρία Λεκόντ. Καλημέρα σας κυρίες και πρόεδρε. Ε, εγώ μένω σε 18 χιλιόμετρα από το αεροδρόμιο Σόλτεγκολ Ρουασί της Γαλλίας. Η κατάσταση είναι απαράδεκτη. Οι πτήσεις ε, μειώνουν το υψόμετρό τους και στις προσγειώσεις και στις απογειώσεις Περισσότερος θόρυβος, περισσότερη χημική μόλυνση, λιγότερος ύπνος, μας λένε σύνεπως ψέματα. Πήρα την απάντηση της κυρίας Ροαγιάλ εδώ και ένα χρόνο. Να σας πω τι πληροφορίες μου δώσανε. Καταρχάς οι χάρτες που στείλανε το Φεβρουάριο του 2014, κυρία Λεκόντ, πρέπει να μιλάτε λίγο πιο αργά. Οι χάρτες λοιπόν που απεστάλησαν το Φεβάριο του 2014 ανταποκρινόντουσαν στις απαιτήσει της οδηγίας 2002-30. Τα ανώτατα όρια θα καθοριστούν από τη Γαλλία και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να παίξει κανένα ρόλο πάνω στο πρόγραμμα δράσης της Γαλλίας. Έτσι μου είπαν πέρυσι. Το πρόγραμμα δράσης αυτό ε, ήταν ακόμα σε επίπεδο προσχεδίου θα έλεγα ο χάρτης του Elden ανταποκρινόταν σε αυτό που ονομάζουμε Elden 56, κάτι το οποίο δεν είναι ε, συμβατό με το πλαίσιο του προγράμματος το οποίο παραπέμπει στο Elden 55. Έχουμε να κάνουμε με 620 ε, με 680.000 κινήσεις, έτσι προβλέπονται για το 2025 ενώ το 2012 είχαμε 497.000 κινήσεις και υπερπτήσεις. Διερωτώμε λοιπόν για τις δυνατότητες δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επιστολή της κυρίας Ρογιάλ μας λέγει ότι θα υπάρξει μία μεταφορά του σχεδίου για το Ρουασία τον αρμόδιο οργανισμό. Πρέπει να γνωρίζει κανείς ότι η διαβούλευση η δημόσια δυστυχώς δεν είναι παρά ένα άλοθη όλα συμβαίνουν έτσι ώστε να μην καταστεί προσβάσιμη για τον πληθυσμό. Εσείς παίρνετε το σχέδιο δράσης για το ΡΟΑΣΥ με τις λεπτομέρειες και τα μέτρα, ενώ ταυτόχρονα εξελίσσεται η ε, διαβούλευση δημόσια. Κάποιοι όμως τοπικοί άρχοντες αποφασίσουν ότι όλα είναι προαποφασισμένα και το καταγγέλουν. Έτσι και αλλιώς για τις ζώνες συγκεκριμένου θορύβου λαμβάνονται κάποια μέτρα, τα λεγόμενα σονοπόντ, τα οποία εγκαθίσταται σε δημόσιους χώρους. Τα αποτελέσματα δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικά και ξέρουν πολύ καλά οι τοπικοί άρχοντες στις περιοχές τους το τι ακριβώς συμβαίνει. Ε, έτσι και αλλιώς οι μαθηματικές ρυθμίσεις οι οποίες γίνονται εκ των υστέρων ε, δεν ε, θα έλεγα ε, δεν έχουν βοηθήσει πολύ τα αεροπλάνα που μας ξυπνούν ξαφνικά στις 2 η ώρα το πρωί. Και εκεί τελειώνει η νύχτα για πάρα πολλούς. Η ADVOCNAR που είναι η Ένωση Άμυνας των κατοίκων των περιοχών αυτών έχει αναγνωριστεί σαν σύλλογος κοινού συμφέροντος. Υπάρχουν ε, ε, περιοχές γύρω από το Ρουασί οι οποίες ε, χαρακτηρίζονται θα έλεγα τα σημεία τα οποία θίγονται περισσότερο από οιαδήποτε άλλα. Η λεπτομερής ανάλυση μας δείχνει ότι οι προτάσεις της γαλλικής κυβέρνησης δεν βρίσκονται στο ύψος των περιστάσεων. Τα μέτρα αυτά είτε είναι εκτός θέματος είτε είναι ασύμβατα με το πνεύμα της οδηγίας 49 των οποίων οι στόχοι είναι υπολογισμός, πρόληψη και μείωση του θορύβου στο εξωτερικό περιβάλλον και όχι στο εσωτερικό περιβάλλον. Πρέπει να ελέγξουμε την χωροτακτική δράση γύρω από το αεροδρόμιο. Κανένας από τους στόχους αυτούς δεν έχει επιτευχθεί. Πρέπει να συνεχίσουμε επίσης την αντιμετώπιση του θορύβου και με μέτρα, με τις μονώσεις ή από το 2015 όμως δυστυχώς ε, ε, έχει διακοπεί η φορολογική διευκόλυνση για τις εργασίες ε, ηχομόνωσης και το πρόγραμμα του 2013 δυστυχώς δεν έχει βοηθηθεί σε τίποτα. Τα μέτρα αυτά είναι και εκτός θέματος, δεν υπολογίζουν και δεν μειώνουν τον θόρυβο στο εξωτερικό περιβάλλον γιατί για, τον, για το εξωτερικό περιβάλλον μιλάει η οδηγία 2249. Θα πρέπει επίσης να απαγορευτούν τα αεροσκάφη χαμηλών επιδόσεων ακουστικά ιδιαίτερα τη νύχτα. Ε, από το 2012 και το 2014 πολλά ε, υπόθηκαν, τίποτα δεν έγινε. Πρέπει επίσης να αναπτυχθούν διαδικασίες πτήσης με μικρότερο θόρυβο. Ήδη αυτό ξεκίνησε το 2012, μειώθηκε ο θόρυβος πολύ λιγότερο από ό,τι είχε αναγγελθεί. Δεν περιμένουμε τίποτα για τα επόμενα χρόνια. Επίσης ε, ε, δημιουργία των λεγόμενων ε, συνεχών διαδικασιών απώλειας ύψους προς προσγείωση. Τίποτα δεν έχει γίνει. Αυτό πάντα βρισκόμαστε στο LDN 55. Δεν έχει υπάρξει καμία αξιολόγηση των μέτρων αυτών σε σχέση με τη μείωση του θορύβου. Συνεπώς λοιπόν εκτός θέματος και αυτό. Κυρία Λεκόντ, να σας ζητήσω να κλείσετε κάπως ε, την συζήτησή σας γιατί κάθε μέλος, ε, ε, κάθε προσκεκλημένος έχει έτσι και αλλιώς μια συγκεκριμένη ομιλία να κάνει. Λοιπόν, το να δημιουργηθεί ένα νέο δίκτυο ε, δρομολογίων μετά την απογείωση από το 2012 δεν έχει δώσει τίποτα. Δεν υπάρχει βούληση της γαλλικής κυβέρνησης. Το ίδιο επίσης και για την ε, απογείωση στο τέλος του αεροδιαδρόμου. Αυτό υποτίθεται ότι εφαρμόστηκε από το 2006 και μετά για το 25% των των απογειώσεων, ανάπτυξη επίσης του δικτύου της παρακολούθησης του θορύβου. Αυτό είναι ενδιαφέρον και θα βοηθήσει. Να συνεχίσουμε να δημοσιεύουμε σε αιτήσια βάση ε, τον θόρυβο ε, της πλατφόρμας GNP. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να λειτουργήσει γιατί δεν υπάρχουν διεθνείς δείκτες σχετικά με τα ΕΛΔΕΝ θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τις μελέτες οι οποίες έχουν ξεκινήσει ήδη, δυστυχώς όμως ε, οι εκθέσεις δεν έγιναν δεκτές. Τι θα γίνει λοιπόν τώρα και τα επόμενα πέντε χρόνια. Να προωθηθεί η διαβούλευση. Δεν θα βοηθήσει σε κανένα από τα τρία, ε, από τα τρία πεδία. Δυστυχώς ε, τα μέτρα αυτά είχαν προταθεί αλλά είναι χωρίς αποτέλεσμα. Τι μπορεί να κάνει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, εναντίον όλων αυτών των καταχρήσεων. Μπορούμε να επηρεάσουμε την Επιτροπή. Δεν θα σας διαβάσω το υπόλοιπο κείμενο. Δυστυχώς δεν υπάρχει τίποτα στις προτάσεις για την κατάσταση η οποία συνεχώς χειροτερεύει. Σας ευχαριστούμε λέει η Πρόεδρος. Ανοίγει τώρα συζήτηση. Ο κύριος Λαβρίο Πρόεδρος, παρακαλώ. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Πρέπει να δώσω πρώτα το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με συγχωρείτε που σας, δια... σας διακόπτω κύριε Λαβρίο. Κανένας δεν ξέρει ποτέ σε αυτό το κοινοβούλιο Μπορεί να, να βρεθεί κανείς σε πολύ δύσκολες καταστάσεις, αλλά δεν θα ήθελα να βρίσκομαι σε αυτή τη θέση. Δίνω το λόγο λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Πάρα πολύ σύντομα. Παρακολουθούμε την κατάσταση, οπότε Ακόμη λαμβάνουμε πληροφορίες, εξ όσων γνωρίζουμε δεν υπάρχει σχέδιο δράσης ε, για το Charles de Gaulle, ε, το αεροδρόμιο του Παρισιού και όσον αφορά τη μελέτη ε, για τις υπερβάσεις του LDN υπήρξαν κάποιες εμπεριστατωμένες γνωμοδοτήσεις ότι για παράδειγμα οι υπερβάσεις έλαβαν χώρα για περισσότερες μέρες από αυτές που επιτρέπονταν αλλά αυτό πρέπει να το ελέγξουμε. Ευχαριστώ πολύ. Μεσή Λαβιό, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. είναι το πρώτο θέμα αντικείμενο αναφοράς από τότε που εξελέγει και είμαι μέλος Επιτροπής εδώ και ένα χρόνο. Είναι παραδεκτή από το 2009. Έξι χρόνια έχουν περάσει που ε, κάθε χρονιά ασχολούμαστε με το θέμα αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία μόλις πήρε το λόγο, ε, πραγματικά ε, είναι πάρα πολύ ε, καλοσυνάτη με την Γαλλία. Αυτό που διαπιστώνουμε όμως ότι καμία από τις δεσμεύσεις της δεν τηρεί η Γαλλία. Όσον αφορά για παράδειγμα το περιβαλλοντικό θόρυβο, η τελευταία επιστολή την οποία πρέπει να λάβατε στις 30 Μαρτίου του 2015, διαπιστώνουμε ότι η Γαλλία ενημέρωσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Νοέμβριο του 2013 ότι υπάρχει ένα σχέδιο δράσης που ε, είχε επεξεργαστεί η Γαλλία για το Charles de Gaulle ε, και το 2013 υποτίθεται ότι είχε δρομολογηθεί. Μέσα Φεβρουαρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακόμη δεν έχει λάβει το σχέδιο δράσης. Υπάρχει ένα θέμα ικανότητας ε, ε, στη γαλλική αρμόδια αρχή. Εν πάση περιπτώσει επίτηδες προσπαθούμε να καθυστερήσουμε το θέμα. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα το οποίο αναφέρθηκε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε ότι 139 υπερβάσεις της ημερήσιας οριακής τιμής ε, διαπιστώθηκαν, ε, ενώ η πρόβλεψη είναι για 35 ημέρες. Εγώ δεν είμαι εμπειρογνώμονας Επιτροπής ε, Περιβάλλοντος, είμαι στην ίδια θέση με τη συνάδελφο Βαλέσα. Δεν ξέρω κατά πόσο η δράση μας είναι η, οδηγία μας είναι ή όχι η σωστή. Ε, πάντως πρέπει η νομοθεσία να γίνεται σεβαστή. Πρώτον, κατά τη γνώμη μου, ε, για το θέμα του περιβαλλοντικού θορύβου κολυσιεργεί η Γαλλία δεν αποφασίζει να ε, έχει, να, να μας παρέχει κάποια κείμενα στα οποία να μπορούμε να βασιστούμε και να επιχειρηματολογήσουμε και όσον αφορά ε, το, την ε, ε ρήπανση του ατμοσφαιρικού αέρα θα ήθελα η Επιτροπή μας να είναι κατηγορηματική ε, απέναντι στη Γαλλία αλλά και απέναντι ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να αναλάβει δράση κατά της Γαλλίας και να ε, καρποφορήσει επιτέλους αυτή η προσπάθεια και να μην χρειάζεται του χρόνου και του παραχρόνου και τρία χρόνια μετά να κάνουμε πάλι την ίδια διαπίστωση γιατί πραγματικά δεν ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσει των πολιτών μας σε κανένα επίπεδο. Ελεονόρα. Θα συμφωνήσω με αυτά τα οποία είπε ο συνάδελφος και να προσθέσω το εξής. Έχω την αίσθηση ιδιαίτερα όταν μιλάμε για διαδικασίες επί παραβάση και ιδιαίτερα τις παραβάσεις τις σχετικές με την ατμοσφαιρική μόλυνση φαίνεται ότι υπάρχει ένα χορός ανάμεσα σε ένα ταγκό ανάμεσα στο κράτος μέλος, τις τοπικές αρχές φτιάχνουν προγράμματα, τα προγράμματα αυτά δεν γίνονται σεβαστά ή δεν εφαρμόζονται εν πάση περιπτώσει, τα όρια ξεπερνιούνται και η διαδικασία αυτή συνεχίζεται από χρόνο σε χρόνο και δεν καταλήγει πουθενά. Ο τομέας αυτός ε, ε, είναι ένα τομέα στον οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει ιδιαίτερα η ατμοσφαιρική μόλυνση. Αλλά δυστυχώς, όπως και στην περίπτωση της Volkswagen, ξέρουμε ότι πολλές φορές οι κανόνες υπάρχουν και εμείς υποτίθεται ότι είμαστε συν, συναποφασίζουμε, είμαστε συνομοθέτες, αλλά δυστυχώς η διαφορά ανάμεσα στη θεωρία και στην πρακτική είναι αβυσαλαία και δεν εφαρμόζονται ποτέ οι ρυθμίσεις αυτές τις οποίες εμείς επιθυμούσαμε να προωθήσουμε. Δεν ξέρω αν θέλει κάποιος άλλος το λόγο. Καλώς σας ευχαριστώ. Αν κατάλαβα καλά λοιπόν. Εμείς θα πρέπει να κρατήσουμε το συγκεκριμένο θέμα ανοιχτό. Στείλαμε μια επιστολή πριν λίγο καιρό στις γαλλικές αρχές. Η απάντηση δεν ήταν ικανοποιητική από πλευρά των γαλλικών αρχών και σε σχέση με το πρόγραμμα δράσης γύρω από το Charles από το αεροδρόμιο Charles de Πρέπει λοιπόν να προχωρήσουν τα προγράμματα αυτά. Δεν είναι δυνατόν να παραμείνουμε ε, στην έλλειψη απάντησης όπως τώρα. Εμείς δεν θέλουμε να δημιουργηθεί μια κατάσταση με προσφυγές από επιπαραλήψεις στη συγκεκριμένη περίπτωση. Θα πρέπει να υπάρξει εν πάση περιπτώσει απάντηση στις ερωτήσεις που έχουν τεθεί. Κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει, αυτή είναι η πρόταση. Οι συνάδελφοι έπρεπε να επιστρέψουν στις πατρίδες τους, δεν είναι εδώ για να τα αποφασίσουν. Θα επιστρέψουμε τώρα στην, στην αναφορά 14, 13, συγγνώμη. 1738 του 13. από την Ένωση εναντίον της α, ανάπτυξης του αεροδρομίου της Σιένα και στις νυχτερινές πτήσεις στο αεροδρόμιο της Σιένα. Υπάρχουν κοινοτικές ρυθμίσεις για την προστασία των πολιτών. Ο αναφερόμενος δεν είναι εδώ, αλλά η Ευρωπαϊκή είναι εδώ και θα της δώσω το λόγο αμέσως. Δεν έχουμε τίποτα να προσθέσουμε σε αυτό το θέμα. Η Σιένα βρίσκεται εκτός αρμοδιότητας αυτής της οδηγίας ούτως ή άλλως. Το αεροδρόμιο της βρίσκεται βρίσκεται εκτός της αρμοδι... του πεδίου αρμοδιοτήτων αυτής της οδηγίας ούτως ή άλλως. There is also a Belgian one. Υπάρχει και μια βελγική αναφορά πάλι του ίδιου ετού για την πανευρωπαϊκή απαγόρευση νυχτερινών πτήσεων πανενοσιακά. Θα θέλατε να λάβετε τον λόγο από αυτού. Δεν είσαστε υποχρεωμένοι να το κάνετε. Μπορείτε να το κάνετε, είναι στη διακριτική σας ευχαίρεια. Ήδη τοποθετηθήκαμε, εντάξει. Πρόεδρος, εντάξει, αρχίζει τώρα ο διάλογος με τους ευρωβουλευτές. Η παρέμβαση των ευρωβουλευτών δεν είναι τόσο πολύ στην αίθουσα αυτή τη στιγμή. Όμως, όμως παρακαλώ, Βοηθήστε με για να συνεχίσουμε με τις αναφορές. Δεν μπορώ μόνοι μου να τα καταφέρω όλα. Λοιπόν, κι άλλο μέλος ευπρόσδεκτο είναι πέμπτη απόγευμα και πολλοί επιστρέφουν στις χώρες τους, στα κράτη-μέλη τους. Και πολλοί από αυτούς, αν όχι περισσότεροι, αεροπορικά. Και δεν πρόκειται για νυχτερινή πτήση, αλλά απογευματινή πτήση και γι' αυτό απουσιάζουν συνάδελφοι. Λοιπόν, αρχίζουν οι παρεμβάσει ευρωβουλευτών. Ποιο ξεκινά. Είναι το 13 λοιπόν. Αναφορά υπαριθμών 13. Εντάξει, αν δεν υπάρχει κανείς που θα ήθελε να παρέμβει, προτείνω το εξή. Λοιπόν, να αποσταλεί μια επιστολή στην Επιτροπή Μεταφορών και Περιβάλλοντος, ΕΝΒΙ και ΤΡΑΝ. Α, όχι για αυτήν, έτσι. Ωραία. Λοιπόν, θα αποστείλουμε μια επιστολή ενημερωτική προς τις δύο κοινοβουλευτικές επιτροπές και κλείνει η αναφορά αυτή. Λοιπόν, γιατί τι μπορούμε να κάνουμε. Ακούσαμε ειλικρινά τοποθετήθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η φυστάμενη νομοθεσία και η οδηγία που ε, βρίσκεται εν ισχύ δεν ασχολούνται με το αεροδρόμιο, με το αερολιμένα Σιένα. Θα έχετε την ευκαιρία να, γίνεται, στην αναφερθείτε στη σύνοψη. Περνάμε στο 16. Αναφορά 0169-2007 κατά των υπερπτήσεων πάνω από πόλεις. Εδώ αφορά τον λιμένα, αερολιμένα Μπαράχα της Μαδρίτης και μια οικιστική περιοχή και την ηχητική ρήπανση και όχληση όσον αφορά την ε, περιοχή αυτή ε, βόρεια της ε, Μαδρίτης ο αναφερόμενος δεν είναι παρόν. Θα ήθελε η Επιτροπή να τοποθετηθεί σε σχέση με το κολμένα Βιέχο στη Μαδρίτη. Σύντομα. Δεν έχει αλλάξει η κατάσταση. Η απάντηση είναι παρόμοια όπως και για τον αερολιμένα Σαρντεγκόρ Βουασί. <clears throat> Αναμένουμε από τις αρμόδιες αρχές να λάβουμε το πρόγραμμα δράσης. Αφορά και τα δύο αυτά θέματα των αναφορών και την Μαδρίτη Μπαράχασα και το Κολμένα Βιέχο. Για την Μπαράχασα μια πρώτη ανάλυση της περίπτωσης δείχνει ότι πρόκειται για τη διαχείριση πτήσεων, <clears throat> υπερπτήσεων και τις δράσεις που περιορίζουν την χρήση του εναέριου χώρου που δεν ρυθμίζεται σε σχέση με τον αντίστοιχο κανονισμό του 2014. Πρόεδρος, πολύ καλά. Εντάξει, λοιπόν, η πρότασή μου γι' αυτό είναι να αναμείνουμε να υποβληθούν περισσότερες πληροφορίες από τις Ισπανικές αρχές <clears throat> που θα αποσταλούν φυσικά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την εφαρμογή του κανονισμού για τους όρους και συνθήκες και ρυθμιστικές διατάξεις και θα επανέλθει στη Γραμματεία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα ενημερώσει μόλις θα έχει ενημερωθεί από τις Ισπανικές Αρχές. Εντάξει, μπορούμε να το κάνουμε αυτό πολύ καλά. Προχωράμε λοιπόν επιτέλους. Πάμε στο 17. Πρόκειται για την αναφορα 17.07.2014. 1707-2014 εξ ονόματος της Ένωσης Κολονιόλα for its future, Κολονιόλα για το μέλλον της και για τις περιβαλλοντικές παραβάσεις στον αερολιμένα όριο Αλσέριο στο Μπέργαμο της Ιταλίας και αναφορά 18-13 του 2014 πάλι για το ίδιο θέμα. Είναι παρούσα η αναφερομένη, είναι η ε, κυρία που έχει τώρα τον λόγο. Παρακαλώ, έχετε τον λόγο κυρία. In qualità di ευχαριστώ Θέλω να ευχαριστήσω την Επιτροπή σας γιατί μας δίνει τη δυνατότητα να σας εκθέσουμε την περίπτωσή μας. Ο σύλλογος μας στράφηκε προς την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί οι Ιταλικοί θεσμοί δεν μπόρεσαν να προστατεύσουν τους κατοίκους της περιοχής. Εμείς ζητάμε τον σεβασμό των κανόνων. Ένα μεγάλο κομμάτι του Μπέργαμο, 7.000 κάτοικοι, 5 σχολεία, 2.000 μαθητές Είμαστε όμοιροι ενός αεροδρομίου το οποίο μεγάλωσε περισσότερο από όσο επιτρεπόταν. Η ανεξέλεγκτη αυτή αύξηση της επιφάνειας του αεροδρομίου συνδέεται με τις πτήσεις Ryanair που αντιπροσωπεύουν το 80% των πτήσεων. Ε, είναι υπό ανάκριση η εταιρεία αυτή στον Πέργαμο για φορολογικές παραδάσεις και έχει τύχει διευκολύνσεων φορολογικών και επιδοτήσεων στο παρελθόν και αυτό το είχε πει και η δήμαρχος της πόλης εκείνη την εποχή. Οι διαχειριστές του αεροδρομίου ελέγχονται κυρίως από τον δημόσιο τομέα και γι' αυτό ακριβώς αυτές οι επιδοτήσεις μπορεί να θεωρηθούν ως παράνομες κρατικές επιδοτήσεις. Ήδη από το 2003 είχε επιτραπεί η αύξηση των δραστηριοτήτων του αεροδρομίου εφόσον μπορούσε να ισορροπηθεί σωστά ο σεβασμός της ε, περιοχής και του αεροδρομίου, το οποίο είναι 3 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης και 2 χιλιόμετρα από την δική μας περιοχή. Δυστυχώς όλα αυτά τα μέτρα αγνοήθηκαν. Το 2015 θα φτάσουμε τις 80.000 κινήσεις αεροπροσγειώσεις το χρόνο και έχει αυξηθεί πάρα πολύ και ο αριθμός των επιβατών. Θα φτάσουμε περίπου στα 10 εκατομμύρια κατέτος επιβάτες. Συνολικά εμπορεύματα και επιβάτες ήταν 6.750.000 ε, όπως ακριβώς φαίνεται και στα στοιχεία του Υπουργείου. Η αδειοδότηση προέβλεπε ότι οι αερομεταφορές θα έπρεπε να αναπτυχθούν προς Ανατολά σε λιγότερο κατοικημένες περιοχές και όχι δυτικά προς την πόλη. Η περιοχή μας δεν έπρεπε να είναι αντικείμενο υπέρπτυσης. Αλλά δυστυχώς όμως ε, ε, πηγαίνουν οι απογειώσεις συνεχώς προς τη Δύση. Από το 2009 και μετά, χωρίς καμία διαβούλευση με τους κατοίκους, υπάρχουν υπερπτήσεις εν στροφή και ε, σε χαμηλό υψόμετρο και αυτό είναι τεράστιο ο κίνδυνος για τους 7.000 κατοίκους και τα 2.000 μαθητές και ξέρετε ότι απαγορεύεται τα σχολεία να είναι κάτω από τους διαδρόμους, ε, από, τις, την πορεία απογείωσης και προσγείωσης των αεροσκαφών. Και ταυτόχρονα παράνομα θα έλεγα η μοναδική περιοχή του Μπέργαμο η οποία ήταν περιοχή κατοικίας με 55 δεσιμπέλ όριο σε μια ζώνη απλού σεβασμού που μπορεί να φτάσει κανείς τα 70 δεσιμπέλ. Όλα αυτά αποφασίστηκαν χωρίς να υπάρξει καμία διαβούλευση εις εναντίον όλων των ρυθμίσεων και Ιταλικών και Ευρωπαϊκών που προβλέπουν τη συμμετοχή των πολιτών σε συγκεκριμένου τύπου επιλογές που έχουν περιβαλλοντική επίπτωση. Η εισαγγελία του Μπέργαμο έθεσε στο αρχείο την αναφορά μας. Έχουμε προχωρήσει σε δύο εφέσεις στο Κεντρικό Δικαστήριο στη Λομβαρδία και στο Συμβούλιο Επικρατείας που ε, κατήργησαν την ζωνοποίηση γύρω από το, αεροσκάφο, από το αεροδρόμιο, αλλά παρόλα αυτά δυστυχώς ε, η περιοχή μας ε, εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προβλήματα με την υπέρπτυση των αεροσκαφών με όρια θορύβου τέσσερις φορές ανώτερα από τα επιτρεπόμενα. Έτσι και αλλιώ τα μηχανήματα παρακολούθησης του θορύβου δεν είναι σε θέσεις οι οποίες είναι κατάλληλες και από τα δεδομένα τους ε, ε, γίνονται επεξεργασίες στοιχείων από την ίδια εταιρεία που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο. Δηλαδή ο ελεγχόμενος είναι ελεκτής του εαυτού του. Ήδη από τον Ιούλιο του 2015 τα πράγματα αλλάξαν διότι η ΕΝΑΚ, η υπεύθυνη για το αεροδρόμιο, απέριψε την δυνατότητα διαφοροποίησης των προσγειώσεων και απογειώσεων χωρίς να δώσει την δυνατότητα στους πολίτες της περιοχής να εκφράσουν την άποψή τους. Εμείς ευχόμεθα η Ευρώπη να επιβεβαιώσει τις βασικές αξίες της προστασίας του περιβάλλοντος και της προστασίας της δημόσιας υγείας. Δεν θα πρέπει να πέσουν θύματα σε οικονομικά συμφέροντα, ιδιαίτερα όταν τέτοια συμφέροντα ε, λειτουργούν με στρεβλό τρόπο στις αγορές. Thank you very much. Σας ευχαριστούμε πολύ και για το ότι συμμετείχατε σε αυτή τη συζήτηση. Η Επιτροπή είναι ελεύθερη να συμμετάσχει στη συζήτηση. Έχετε τον λόγο αν επιθυμείτε να παρέμβετε. Μια και από πλευρά αναφερομένου έχει αναφερθεί ένα διαφορετικό σημείο, θα ήθελα να διευκρινίσω κάτι σε σχέση με την οδηγία του, την αντίστοιχη οδηγία του που ρυθμίζει αυτόν τον τομέα. Αν η αύξηση στις ενέργειε μεταφορές ή η αλλαγή απογειώσεων, τροποποίηση απογειώσεων ή τα αεροπλάνα δεν συνεπάγονται κάποια νέα εργοτάξια ή νέα διεύρυνση αεροδρομίων στην χερσαία περιοχή, οι αλλαγές αυτές των αερολιμένων δεν εντάσσονται στο πλαίσιο της οδηγίας της ΑΕΚΑΟ. Δεν δηλαδή απαιτούν μια αξιολόγηση, εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Δεν απαιτείται κάτι τέτοιο. Όσον αφορά την οδηγία 2001-42, όπως από πλευράς αναφερομένου σωστά ε, τονίζεται, αυτή η ε, ακουστική, ηχητική επίπτωση και η ρύθμιση μπορεί να θεωρηθεί ένα ε, πρόγραμμα που θα εντασσόταν σε αυτή την οδηγία μια και όμως αυτός ο ακουστικός χάρτης η, η ε, από το τοπικό δικαστήριο και η νομολογία αυτή επιβεβαιώθηκε και από το ε, πρωτοδικείο μετά δεν υπάρχει καμιά ανάγκη να αναλυφθεί οποιαδήποτε πρωτοβουλία ή δράση, μια και οι εθνικές αρχές ήδη δραστηριοποιήθηκαν και ανέλαβαν δράση σχετικά. Όσον αφορά με την οδηγία του 2002-49, ε, μπορεί να ενημερωθεί ο αναφερόμενος ότι έχει ασκηθεί ήδη διαδικασία προσφυγή επί κατά της Ιταλίας όσον αφορά την έλλειψη προσαρμογών σε σχέση με τα προγράμματα, με πρόγραμμα δράσης και το αεροδρόμιο του Μπέργαμο καλύπτεται από αυτή την προσφυγή. Όσον αφορά την ρήπανση του ατμοσφαιρικού αέρα και σε σχέση με την οδηγία 2008-50 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ξεκίνησε μια διαδικασία επί παραβάση όσον αφορά το υπερβολικό ποσοστό ε, οξυδίων του αζότου στην ατμόσφαιρα και καλύπτεται και το αεροδρόμιο του Μπέργαμο σχετικά με αυτή την προσφυγή. Επίσης θα ήθελα να αναφέρω ότι επίσης ερεύνησε η Επιτροπή τα σχετικά με την ε, υπέρβαση στα PM10 μικροσωματίδια και έτσι και το Μπέργαμο καλύπτεται και από αυτή την πτυχή ως αεροδρόμιο. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, λοιπόν, όπως βλέπετε, καμιά φορά κινούνται τα πράγματα και κινούνται και αρκετά γοργά κιόλα. Έχουμε λοιπόν δύο διαδικασίες επί παραβάση κατά της Ιταλίας σε σχέση με αυτό το θέμα. Με άλλα λόγια, δύο μ, υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον του δικαστηρίου. Δηλαδή θα παραμείνουν ανοιχτές αυτές οι αναφορές μέχρι ότου υπάρχει, υπάρχει νομολογία, απόφαση δικαστηρίου. Και θα ενημερωθεί κιόλα ε, και αν αυτό είναι βούληση των μελών τη Επιτροπή, μπορεί να αποσταλεί μια επιστολή προ τη μόνιμη αντιπροσωπεία τη Ιταλία στι Βρυξέλλες ότι παρακολουθούμε αυτή την περίπτωση εκ του σύνεγγυ προσεκτικά και αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει σε σχέση με την έκβαση των προσφυγών που έχουν ασκηθεί κατά της Ιταλίας. Αυτό είναι αυτό που μπορούμε ουσιαστικά να πράξουμε και αυτό θα κάνουμε. Θα λάβει τώρα τον λόγο η κυρία Καρτίνη και μετά μπορούμε ίσως να ολοκληρώσουμε επ' αυτού. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να προσθέσω μόνο μία πληροφορία αν επιτρέπετε. Ίσως αφορά τώρα και ποιες είναι οι προσδοκίες ε, ε, των εκπροσώπων των πολιτών ε, σε σχέση με αυτά τα θέματα. Υπάρχει ένα νέο πρόγραμμα ανάπτυξης και δράσης το οποίο πρόκειται να ληφθεί υπόψη. Και έτσι λοιπόν σύντομα θα έχουμε νέες εκτιμήσεις που θα γίνουν και όλα αυτά θα επικαιροποιηθούν με νέα στοιχεία τα οποία θα ε, κατατεθούν και ελπίζουμε ότι έτσι θα μπορέσουμε να βρούμε μια διέξοδο από αυτό το αδιέξοδο ε, το οποίο δημιουργεί και μια απεσιοδοξία ίσως. Λοιπόν, επ' αυτού ζητήθηκε ίσως αν μπορούμε να πούμε δύο λόγια επ' αυτού. Δηλαδή ουσιαστικά ανέφερα ότι σύντομα θα έχουμε αυτό το πρόγραμμα, αναπτυξιακό πρόγραμμα, το οποίο θα κατατεθεί και θα υπάρξει μια νέα μελέτη επιπτώσεων και βιωσιμότητας. Το χαιρετίζουμε αυτό σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές και ιταλικές ε, διατάξεις, ίσως θα μπορούσε το ένα ή το άλλο να μπορέσει να διευθετηθεί. Όμως υπάρχει κάποια απεσιοδοξία και ήθελα να δούμε τι μπορούμε να ακούσουμε και να πούμε. Πρόεδρος. Λοιπόν, σημειώσαμε προσεκτικά αυτά τα οποία μας είπατε. Θα συμπεριληφθούν στην επιστολή που θα αποστείλουμε στις Ιταλικές Αρχές. Ίσως αυτό θα αυξήσει την πίεση κάπως περισσότερο από πλευράς μας έναντι των Ιταλικών αρχών. Βλέπω λοιπόν συμφωνείτε μαζί μου επί της ουσίας επ' αυτού του θέματος. Συμφωνούμε να κάνουμε αυτό. Πολύ καλά, εξαιρετικά λοιπόν. Αυτό θα πράξουμε. Φυσικά είναι μια εκκρεμούσα περίπτωση δικαστικά, θα παραμείνει ανοιχτή αναφορά μια και ακόμα εκκρεμεί η δικαστική, η δικαστική εξέταση. Και θα προσεγγίσουμε, θα αποστείλουμε αυτή την επιστολή στις Ιταλικές Αρχές λέγοντας ότι η Επιτροπή Αναφορών παρακολουθεί του σύνεγγυς τα όσα συμβαίνουν σε αυτού του ε, θέματος στην Ιταλία. Περνάμε στην επόμενη αναφορά που είναι η ε, αναφορά 0112-2015 του Ρομπέρτο, Μπαρκαρόλη σε σχέση με τη ρήπανση που προκαλείται από την εναέρια κυκλοφορία από και προς τα αερολιμένα Τσαμπίνο στη Ρώμη. Ο κύριος Μπαρκαρόλη είναι παρόν. Με χαρά του δίνω τον λόγο. Παρακαλώ κύριε Μπαρκαρόλη. Um, Έχω κάποιες διαφάνειες. Parlo anche senza slide. E, intanto Αλλιώς μπορώ και να μην τις χρησιμοποιήσω. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι το αεροδρόμιο Τσαμπίνο εγώ εκπροσωπώ εδώ την Επιτροπή για τη Μείωση Περιβαλλοντικού Αντικτύπου του Αερολιμένου Τσαμπίνο επίσημες είναι οι πτήσεις που γίνονται ε, και οι προσγειώσεις και οι απογειώσεις στο Τσαμπίνο εδώ και 13 χρόνια έχει δημιουργήσει μια εναέρια κυκλοφορία από το 2002 και μετά πάρα πολύ σημαντική. Και η... καμία από τις σχετικές οδηγίες δεν έχει γίνει ε, σεβαστή, ούτε, ούτε η περιφαλλοντική νομοθεσία, ούτε η νομοθεσία για την ηχορύπανση. Το αεροδρόμιο Τσαμπίνο είναι ένα από τα παλαιότερα αεροδρόμια ε, στον κόσμο. Κάποτε είχε πάρα πολύ λίγους ε, επιβάτες ε, κατ' Έχουμε περάσει σε Έχουμε περάσει από ένα εκατομμύριο επιβάτες κατέτος σε πέντε εκατομμύρια κατέτος. Ε, το Τσαμπίνο δεν κάνει μόνο επιβατικές μεταφορές αλλά ε, και ε, πολιτική αεροπορία γενικότερα, στρατιωτικές πτήσεις επίσης και όλες αυτές οι πτήσεις προσγειώνονται και απογειώνονται σε 150 μέτρα από πολυκατοικίε τη πόλη του Τσαμπίνο. Εκεί τελειώνει το αεροδρόμιο, στα 150 μέτρα από σπίτια. Και αυτό ίσχυε πάντα, 100 χρόνια είναι έτσι η κατάσταση. Η πόλη Τσαμπίνο είναι 150 μέτρα δίπλα στον αεροδιάδρομο. Ε, υπάρχουν πολύ χαμηλές υπερπτήσεις ε, του περιφερειακού του πάρκου του Λάμπη Αντίκα, που είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πάρκο από ιστορικής και περιβαλλοντικής απόψεως ε, είναι κοντά στο Τσαμπίνο και γίνονται υπερπτήσεις κατά τις απογειώσεις και τις προσγειώσεις. Ένα τμήμα του νοτίου της Ρώμης όπου 400.000 ε, άνθρωποι διαμένουν. Γίνονται λοιπόν υπερπτήσει του Τσαμπίνο αλλά και, τη, και της ε, κοινότητας Μαρίνο ε, όπου διαβιούν 4.000 άτομα ζητήσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, ξεκινήσει διαδικασία επί παραβάση. Έχει ξεκινήσει αυτή η διαδικασία, ε, μια διαδικασία EU Pilot όσον αφορά τον αερολιμένα Τσαμπίνο ε, στη Ρώμη. ε, υπήρξε μάλιστα δέσμευση από τους εκπροσώπους του αερολιμένα επί συγκεκριμένων σημείων πρώτον να γίνουν εκ των υστέρων ε, αξιολογήσεις περιβαλλοντικού αντικτύπου μετά από το 2002 όπου και σημειώθηκε τεράστια αύξηση σε αέριες κυκλοφορίες όπως επίσης αλλαγές στη διάρθρωση του αερολιμένα ε, που θα έδιναν την δυνατότητα εφαρμογής ε, των σχετικών οδηγιών η Ευρωπαϊκή Ένωση μας είχε πει ότι θα γινόταν, ε, θα υπήρχε ένα γενικό σχέδιο αστικού αερολιμένα με συγκεκριμένους περιορισμούς για περιβαλλοντικούς λόγους και πριν από μερικές ημέρες μόλις ε, η Εθνική Αρχή ξεκίνησε μια διαδικασία περιβαλλοντικής αξιολόγησης ε, βάσει ενός γενικού προγράμματος, ενός γενικού σχεδίου, όμως δεν η, αλλαγή που θα γίνει ότι θα είναι πια διευτερεύον αυτό το αεροδρόμιο το οποίο θα, ε, θα χρειάζεται να συμμορφώνεται με μικρότερες περιβαλλοντικές προδιαγραφές ε, θα είναι μικρότερη δηλαδή η κυκλοφορία. Γίνεται λοιπόν μια αξιολόγηση βάσει μιας πιο περιορισμένης νομοθεσίας ε, και η συμβολή της δημόσιας διαβούλευσης περιορίζεται σε 30 και όχι σε 60 ημέρες. Επίσης, το είδος της περιβαλλοντικής αξιολόγησης που θα γίνει δεν θα είναι ε, πλήρε, θα είναι περιορισμένη η περιβαλλοντική αξιολόγηση λόγω της νομοθεσίας που θα ισχύσει εν προκειμένου είναι ένα από τα τελευταία ψέματα που μας έχουν πει οι εθνικές αρχές όσον αφορά τον αερολιμένα αυτόν. Είχαμε πει ότι θα μπορούσε να γίνει ένας νέος αερολιμένας κάπου αλλού, δηλαδή το τσαμπίνο να αντικατασταθεί ε, στο ρόλο του κάτι το οποίο είχε αποφασιστεί το 2010. Μετά το 2012 όμως είπαμε ότι θα γίνει όταν αναδιάρθρωση και ότι θα πήγαινε η επιπλέον εναέρια κυκλοφορία στο Φιουμιτσίνο. Κάτι το οποίο μπορεί να γίνει αυτή τη χρονιά. Ε, η, ξεκίνησε η διαδικασία της σχετικής οδηγίας, ε, δεν είναι πλέον ένα αεροδρόμιο πόλης, αλλά ένα αεροδρόμιο δευτερεύων, επικουρικό. Ε, θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που παρίσταται σήμερα να μας πει ποια είναι η ε, στάση της έναντι των Ιταλικών αρχών γιατί οι Ιταλικές αρχές πρέπει να σεβαστούν την εθνική νομοθεσία και την ενωσιακή νομοθεσία και πρέπει να εξασφαλίσουν την πρόσβαση του κοινού όπως επίσης και να εξασφαλίσουν την υγεία των πολιτών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μήπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να μας πει ορισμένα πράγματα επ' αυτού. Πράγματι, όπως είπαν και οι αναφερόμενοι έχουμε ξεκινήσει μια διαδικασία. Είναι τρέχουσα η διαδικασία αυτή. Εδώ και λίγες ε, μέρες ξεκίνησε μια νέα διαδικασία του EIA για το νέο master plan της περιοχής. Στις προηγούμενες απαντήσεις τις οποίες σας είχαμε στείλει, οι Ιταλικές αρχές ανέλαβαν την υποχρέωση να εφαρμόσουν τις αποφάσεις του παρελθόντος. Και θα ήθελα εδώ να προσκαλέσω τον αναφερόμενο να υποβάλει όλες τις παρατηρήσεις τις οποίες έκανε σχετικά με το συγκεκριμένο αεροδρόμιο στο Υπουργείο Περιβάλλοντος της χώρας του, διότι όπως είπα έχει ξεκινήσει μια διαδικασία ελέγχου. Η προθεσμία είναι στο τέλος μάλλον στις αρχές Δεκεμβρίου. Η υπεύθυνη για τον έλεγχο επιτόπου είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Να αναφέρω επίσης ότι αυτή η διαδικασία του EIA που βρίσκεται σε εξέλιξη είναι συμβατή με την οδηγία έχει υπάρξει γύρω από το θέμα αυτό στο παρελθόν μία πρόταση προσφυγής επί παραλήψη, αλλά τέθηκε στο αρχή. Γιατί ο Ιταλικός νόμος, ο οποίος επέτρεψε την εφαρμογή της συγκεκριμένης διαδικασίας, είναι συμβατός με την κοινοτική οδηγία. Ένα τελευταίο σημείο τώρα, σχετικά με το θόρυβο. Όπως είπαμε και πριν, έχουμε μια διαδικασία η οποία συνεχίζεται σε σχέση με τη μη εφαρμογή των χαρτών θορύβου και η περίπτωση του αερολιμένα του Τσαμπίνο καλύπτεται. Λοιπόν, η συνάδελφος, η κυρία Εύη. Είναι παράλογο να βλέπει κανείς ότι ένα δημόσιο αεροδρόμιο, ένα κρατικό αεροδρόμιο, το αεροδρόμιο του Τσαμπίνο, έχει λειτουργήσει όλα αυτά τα χρόνια, τα τελευταία 13 χρόνια, χωρίς να έχει υπάρξει ε, μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων ως όφιλε. Έχει λειτουργήσει ε, απολύτως ε, ελεύθερα. Η προστασία του περιβάλλοντος και η προστασία μέσω ακριβώς των ε, συγκεκριμένων μελετών ακολουθεί κάποια μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί για τον έλεγχο της κατάστασης. Εδώ φαίνεται ότι οι προθεσμίες ε, περνούν η μία μετά την άλλη και αυτή τη στιγμή μετά από 13 χρόνια γίνεται μία μελέτη επιπτώσεων Πώς μπορεί κανείς να αξιολογήσει με αντικειμενικότητα την κατάσταση του περιβάλλοντος. Είναι απαραίτητο λοιπόν στην παρούσα φάση να συνεχίσουμε την διαδικασία, αλλά επαναλαμβάνω μου φαίνεται εντελώς παράλογο πως και από πλευράς των κοινοτικών οργάνων δεν έχει υπάρξει έλεγχος των διαδικασιών και του σεβασμού των χρονικών προθεσμιών Εγώ δεν μπαίνω στην ουσία της αξιολόγησης, κατανοώ ότι είναι αρμοδιότητα του κράτους μέλους, αλλά παρόλα αυτά ο χρονισμός των προθεσμιών δηλαδή είναι κάτι το οποίο ενδιαφέρει και την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία πρέπει να απαιτήσει να γίνουν σεβαστοί οι κανόνες. Δεν ξέρω αν υπάρχει εδώ κάποια εκπρόσωπος ε, της Ιταλικής ε, Προεδρίας και αυτό δείχνει ότι η Ιταλία δεν δίνει σημασία στο σεβασμό των ευρωπαϊκών της υποχρεώσεων. Ελπίζω να δραστηριοποιηθεί επιτέλους η Ιταλία έτσι ώστε να προσπαθήσουμε να λύσουμε το συγκεκριμένο πρόβλημα το οποίο θα έλεγα επηρεάζει τόσες πολλές οικογένειες δεν ξέρω αν είδατε καλά την απόσταση που υπάρχει από την κατοικία μέχρι το αεροδρόμιο. Μιλάμε για 150 μέτρα. Πραγματικά κάτι το απαράδεκτο. Στην ουσία είναι ένα αεροδρόμιο μέσα στο μέσο της πόλης. Και σύν της άλλης έχει χτιστεί το αεροδρόμιο δίπλα ακριβώς από το πάρκο της Απιαντίκα Πάρα πολλά θα έπρεπε να προστατεύσουμε ιστορικά μνημεία Και, τα λοιπά και δεν το κάνουμε αυτό. Λοιπόν, ελπίζω να γίνει το ταχύτερο δυνατόν ό,τι χρειάζεται για να πιέσουμε τις Ιταλικές αρχές. Έτσι ώστε από πλευρά τους να πάρουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα και να αναλάβουν δράση. Είστε συνάδελφος. Θα μας πείτε ποιος είστε γιατί δεν είναι το καρτελάκι μπροστά σας. Ναι. Βε, βεβαίως, ο κύριος Νταμπουράνο. Είμαι βουλευτής της Cinque Stelle από την εκλογική περιφέρεια του αναφερομένου. Άκουσα με προσοχή αυτά τα οποία είπε η Εύη, η συνάδελφος Εύη, και να κάνω δύο παρατηρήσεις, μια ειδική και μια γενικότερη. ειδική. Ξέρετε ότι θα γίνει ένα εξαιρετικό ιοβιλέο για την πόλη, στη Ρώμη, και εδώ έχουμε να κάνουμε με σαφέστατη παραβίαση των ε, οδηγιών και δυστυχώς θα υπάρξει μια αύξηση του αριθμού των επιβατών και σε σχέση με τη μόλυνση και σε σχέση με την ηχομόλυνση. Και τώρα μια γενική παρατήρηση. Εδώ μιλάμε για την τελευταία δυνατότητα των κατοίκων είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ο μοναδικός τρόπος που έχουν πλέον για να επιβεβαιώσουν την ορθότητα των θέσεών τους και θα χρησιμοποιηθεί αυτό θα έλεγα για να αποδειχθεί και η χρησιμότητα των ευρωπαϊκών θεσμών γιατί οι Ιταλικές αρχές στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι εκτός ορίου νομιμότητας. Προφανώς και μας ενδιαφέρει, όλοι είμαστε Ευρωπαίοι πολίτες και όλοι ενδιαφερόμεθα για τους υπόλοιπους Ευρωπαίους και όπως είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η συνεχιζόμενη ερευνητική διαδικασία εξελίσσεται. Θέλουμε κάποια ενημέρωση σε σχέση με τις πληροφορίες οι οποίες δόθηκαν πρόσφατα στην Επιτροπή και περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επανέλθει στην γραμματεία της να έρθει σε επαφή δηλαδή με την γραμματεία μας όταν έχει τα νέα στοιχεία και θα ήθελα να επαναλάβω προς τον αναφερόμενο αυτά τα οποία είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι οι παρατηρήσεις σας θα πρέπει να κατατεθούν και στις εθνικές αρχές. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει πολύ. Εφόσον συμφωνούν μαζί μου οι συνάδελφοι, προτιμώ να κρατήσουμε την αναφορά ανοιχτή. Η διαδικασία συνεχίζεται έτσι κι αλλιώς και να στείλουμε μια πολύ σύντομη επιστολή προς τις Ιταλικές αρχές ζητώντας από τις αρχές αυτές να μας δώσουν τις απαιτούμενες διευκρινήσεις. Και επιστέψτε μου συνάδελφοι, έχουν υπάρξει περιπτώσεις στο παρελθόν όπου μια απλή επιστολή από αυτήν την Επιτροπή άλλαξε τα πράγματα. Και δεν το λέω αυτό για να φανώ καλή. Έχει αποδειχθεί ότι ότι το θέμα των απλών επιστολών από πλευράς μας είναι μια μέθοδος αποτελεσματική όταν οι, βασικές, οι τοπικές αρχές βλέπουν ότι ασχολούμεθα με τα θέματα αυτά τότε παίρνουν τα σωστά μέτρα και η επιστολή αυτή φυσικά θα δημοσιοποιηθεί. Λοιπόν, κλείνουμε το θέμα αυτό έτσι όπως είπαμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα έχω πάρα πολλούς αναφερομένους, τους οποίους θα ήθελα να δώσω το λόγο δύο λεπτά στον καθένα. Όχι περισσότερο, γιατί έχουμε τα υπόλοιπα θέματα. Γέγκερ ή ο συνάδελφός σας, όποιος θέλει έχει το λόγο. Λέγομαι Στιούαρτ, είμαι συνάδελφος της Σουζάν. Θέλω να σας ευχαριστήσω που αναφερθήκατε στην αναφορά μας και που μεταφέραμε στις άλλες, μεταφέρατε στις άλλες επιτροπές την αναφορά μας. Υπάρχει ο κίνδυνος κανένας να μην ασχοληθεί με το θέμα της φορολογίας, όπως σωστά είπατε. Ίσως αυτή τη στιγμή να μην παραβιάζονται οι προβλέψεις της οδηγίας, αλλά τα μεμονωμένα κράτη-μέλη είναι ιδιαίτερα διστακτικά στην εφαρμογή φόρων στα καύσιμα των αεροσκαφών, γιατί θεωρούν ότι έτσι οι αερομεταφορεί του θα σταματήσουν να είναι ανταγωνιστικοί. Γι' αυτό λοιπόν εγώ θα ήθελα να κλείσουμε τη συζήτηση λέγοντας ότι υπάρχει κίνδυνος να μην συμβεί τίποτα. Γιατί ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα θεωρήσει ότι είναι δική της ευθύνη, ούτε τα κράτη-μέλη θα πάρουν τα απαιτούμενα μέτρα. 45 δευτερόλεπτα για τη Σουζάν. Δεν ξέρω αν μπορούμε εμείς στο μέλλον να παρακολουθήσουμε τη διαδικασία αυτή, να μην χάσουμε δηλαδή την επαφή με την αναφορά μας. Ίσως αργότερα στο τέλος να μου δώσετε μια συνολική απάντηση. Πέραν τούτου θέλω να σας ευχαριστήσω Είδα ότι παρατηρήσατε το μέγεθος και την κλίμακα του προβλήματος που έχει προκαλέσει ακριβώς και τις πρωτοβουλίες των πολιτών σε όλη την Ευρώπη. Είναι προφανές σήμερα μετά από αυτά που ακούσατε πόσο μεγάλο και σημαντικό είναι. Σας ευχαριστώ. Μπράντε. Όχι. Le Για Η Αντουάν Βιλεμής. Να σας ευχαριστήσω Πρόεδρε, να ευχαριστήσω και την Επιτροπή Αναφορών που κρατάτε ανοιχτή την αναφορά μας, που καταλάβατε το μέγεθος του προβλήματος και που ζητήσατε από το Βέλγιο διευκρινήσεις. Το Βέλγιο είναι μια χώρα που δεν είναι ενιαία ουσιαστικά, είναι τρεις περιφέρειες, αλλά το Ομοσπονδιακό κράτος είναι αυτό το οποίο είναι υπεύθυνο για τον καθορισμό των αεροδιαδρόμων και είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή των κοινοτικών ρυθμίσεων απέναντι στα ευρωπαϊκά όργανα. Τώρα, Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος. Είπατε ότι υπάρχουν πολλές ε, ρυθμίσεις νομοθετικές ευρωπαϊκές. Κατανοούμε τον κανονισμό του, 94, του 2014-987. Αλλά υπάρχει επίσης και ο 249 που επιτρέπει να αναλαμβάνονται και να σχεδιάζονται πρώτα προγράμματα δράσης για την καταπολέμηση του θορύβου. Αυτό δεν έχει προχωρήσει στο Βέλγιο λόγω της φύσης του βελγικού κράτους γιατί τα προγράμματα είναι αντιφατικά μεταξύ τους, καθορίζονται στις περιφέρειες και υπάρχει μια πλήρης έλλειψη ε, αποτελεσματικότητας με αποτέλεσμα να παραβιάζουμε συστηματικά όλους τους κανόνες σωστής ευρωπαϊκής διακυβέρνησης και ορθής πρακτικής, δεν αποφεύγουμε την υπέρπτυση από το κέντρο των πόλεων, της πρωτεύουσα στη συγκεκριμένη περίπτωση, έχουν ξεκινήσει προσφυγές επί παραλήψη και σε άλλα κράτη-μέλη. Είμαστε στην καρδιά των ευρωπαϊκών οργάνων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να ξεκινήσει μια διαδικασία επί παραβάση ε, γιατί δεν εφαρμόζει την οδηγία 2049. Κυρία Λεκόντ, δύο λεπτά. Να σας ευχαριστήσω Βλέπω ότι η Γαλλία για μια ακόμη φορά δεν είναι στο ύψος των περιστάσεων και αυτό επιβεβαιώνει και τον τρόπο που αντιμετώπισαν την αντιπροσωπεία μας την Τρίτη το απόγευμα. Μας δέχθηκαν υπεύθυνοι του Υπουργείου Οικολογικών Υποθέσεων και δεν μας είπαν απολύτως τίποτα. Είπαν ότι θα δουν τα πράγματα και θα κάνουν προτάσεις. Ευχαριστώ. Χαίρομαι που παραμένει ανοιχτή η αναφορά αυτή, ήταν απαραίτητο αυτό και ελπίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει μέτρα απέναντι σε μια κυβέρνηση η οποία αυτή τη στιγμή διαπράττει μια παράβαση. Ευχαριστώ πολύ. Αρτσούφι. Ευχαριστώ. Ένα μέλος της, του συλλόγου, η κυρία Πέσε. Ευχαριστώ. Εμείς θέλουμε να επιβεβαιώσουμε αυτά τα οποία είπε και ο προηγούμενος ομιλητής. Στραφήκαμε στην Ευρώπη γιατί εμείς παρουσιάσαμε τα θέματα μας σε όλα τα ευρωπαϊκά και ιταλικά, στα ιταλικά όργανα. Δεν υπήρξε ανταπόκριση. Υπουργείο Μεταφορών, Υπουργείο Περιβάλλοντος, Προεδρία της Κυβέρνησης, Πρόεδρος της, της Δημοκρατίας. Αυτή τη στιγμή υποστήκαμε τεράστια οικονομικά βάρη για να βγουν αποφάσεις ευνοϊκές για μας, αλλά δεν υπήρξε τίποτα. Φοβόμαστε λοιπόν γιατί μιλάμε για ακόμα μεγαλύτερη μεγέθυνση του αεροδρομίου Όριο Ντισέριο. Εμείς αντίθετα με το Τσαμπίνο έχουμε να κάνουμε με συγκεκριμένα μέτρα τα οποία απλά δεν γίνονται δεκτά. Ξεπερνάμε όλα τα όρια και αναμένεται αύξηση ενός μικρού αεροδρομίου που έχει αποκτήσει τεράστιες διαστάσεις και έχει καταστεί τώρα το τρίτο στην Ιταλία σε κινήσεις. Είναι παράλογη η πραγματικότητα αυτή και αυτό οφείλεται ότι σε 50 χιλιόμετρα <clears throat> βρίσκεται ένα αεροδρόμιο το οποίο δεν χρησιμοποιείται με μηδενικό θα έλεγα έργο και γι' αυτό το λομβαρδικό πρόγραμμα για, τους, για τα αεροδρόμια είναι η μοναδική λύση. Αλλά δυστυχώς αυτό το οποίο γνωρίζουμε σήμερα είναι ότι αν παρέμβει η Ευρωπαϊκή Ένωση κάτι θα συμβεί, γιατί μέχρι τώρα οι παρεμβάσεις μας στις Ιταλικές αρχές δεν έχουν αποδώσει απολύτως τίποτα. Αυτή είναι μια φωνή ενός πραγματικού Ευρωπαίου. Χαίρομαι που σας άκουσα. Καλώς. Κλείνουμε λοιπόν. Λοιπόν, αυτό ολοκληρώνει όλα τα θέματα όσον αφορά τις εναέριες μεταφορές, αεροπορικές εταιρείες, ρήπανση της ατμόσφαιρας. Έχω και άλλο ένα ομιλητή. Ρομπέτο Μπαρκαρόλη. Παρακαλώ κύριε Μπαρκαρόλη, έχετε τον λόγο. Ε, να ευχαριστήσω και εγώ την Επιτροπή σας για το ενδιαφέρον σας και που διατηρείτε ανοιχτή την αναφορά μας. Ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προσπάθεια την οποία έκανε έτσι ώστε να μείνει ανοιχτή και η διαδικασία επί παραβάση η αναπομπή της υπόθεσης στις Ιταλικές αρχές, όπως είπε η συνάδελφος από τον Πέργαμο, δεν είναι κάτι το αποτελεσματικό. Εμείς έχουμε κάνει προσφυγή ε, και στα δικαστήρια καταθέσαμε 1500 καταγγελίες. Αυτό στην Ιταλία όμως δεν είναι αποτελεσματικό. Η διαδικασία η οποία έχει ξεκινήσει από την ΕΝΑΚΑ, από την αρμόδια αρχή για τα αεροδρόμια. Ξεκίνησε μόνο και μόνο γιατί υπάρχει η διαδικασία EUPILOT. Μόνο και μόνο δηλαδή γιατί υπήρξε ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της δικής σας Επιτροπής. Αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εσείς μειώσετε την πίεση προς τις Ιταλικές αρχές, οι Ιταλικές αρχές θα συνεχίσουν να λένε ψέματα. Σας ζητάμε λοιπόν να συνεχίσετε την πίεση γιατί αυτό θα βοηθήσει την Ιταλία να φτάσει τον επιθυμητό ευρωπαϊκό μεσόρο. Μπορώ να σας διασφαλίσω κύριε ότι σημειώσαμε προσεκτικά τις δηλώσεις σας εδώ απόψε. Και μπορώ επίσης να σας διασφαλίσω ότι <clears throat> δεν στραφεί έγινε κάποια παρέμβαση σε εμά στην Επιτροπή Αναφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάταια, επί Ματέο. Πολύ σοβαρά τα λαμβάνουμε όλα αυτά υπόψη, αλλά έχουμε περιορισμένο φάσμα δραστηριοτήτων στο εύρος τους και η αρχή της επικουρικότητας όπως ισχύει η Ευρωπαϊκή Οδηγία κατά τα άλλα πρέπει να μας κάνει να σταθμίσουμε πολύ προσεκτικά το τι μπορεί να γίνει ή όχι. Παρ' όλα αυτά ήταν πολύ σωστό αυτό που κάναμε. Κάναμε, υιοθετήσαμε μια οριζόντια προσέγγιση, ασκήσαμε μια, κάναμε μια πρωτοβουλία ακούσαμε τις παρεμβάσεις σας και εσείς μας βοηθήσατε να δούμε τις διάφορες πτυχές ε, των θεμάτων αναφορών που μας κατατέθηκαν. Η οριζόντια λοιπόν αυτή προσέγγιση επίσης ε, θα υποβληθεί, θα διαβιβαστεί στην Επιτροπή Μεταφορών και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Με μια επιστολή από πλευράς μας που θα τονίζει το μεγάλο ενδιαφέρον που εκφράζουν οι πολίτες μας τον αριθμό εκείνων που εσείς μπορέσατε να συνεκπροσωπήσετε αναλαμβάνοντας αυτή την πρωτοβουλία σας και την ε, περιβαλλοντική, τα περιβαλλοντικά προβλήματα τα οποία μπορούν να συνεπάγονται τέτοιου είδους καταστάσεις και φυσικά το ότι πλήττονται άνθρωποι από όλα αυτά. Αυτό είναι όλο που μπορούμε να κάνουμε. Και με αυτό τώρα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για το ότι προσήλθατε εδώ ταξιδέψατε, καλύψατε μεγάλη απόσταση για να έρθετε στις Βρυξέλλες, έλαμπε ο ήλιος όταν φτάσατε ε, και τώρα άλλαξε ε, αυτός ο όρος. Θα συνεχίσουμε να προσέχουμε, να έχουμε υπόψη το θέμα αυτό το οποίο αναφέρατε. Είσαστε πάντα, έχετε τη δυνατότητα να έρχεστε σε επαφή με τη γραμματεία της Επιτροπής Αναφορών για να δείτε πού βρίσκεται η αναφορά σας, αν υπάρχουν άλλες παρόμοιες αναφορές που έχουν κατατεθεί ή υποβάλλονται κτλ. Να είσαστε λοιπόν πάντα σε επαφή μαζί μας και εμείς θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να είμαστε σε επαφή μαζί σας. Αυτά είναι σημαντικά ενημερωτικά λοιπόν λοιπόν προς όλους σας, ε, για όλους εσάς που εμπλέκεστε σε αυτές τις αναφορές για τα θέματα αερομεταφορών. Σας ευχαριστούμε που προσήλθατε. Καλό ταξίδι επιστροφής στη ε, πατρίδα σας, στη χώρα σας. Σας ευχόμαστε κάθε καλό, κάθε επιτυχία. Προχωρούμε τώρα με αναφορές σε ένα τελείως διαφορετικό ζήτημα. Ένα θέμα όπως ε, την αναφορά 2348 κάθετος 2014 με περιορισμούς όσον αφορά τον πληθυσμό λύκων στη Σαξονία της Γερμανίας. Και υπάρχει και μια άλλη αναφορά, αλλά θα την δούμε ξεχωριστά, μια άλλη αναφορά, θα την δούμε ως ξεχωριστή περίπτωση. Ο κύριος Άντορφ Βίτ είναι παρόν, έχει τον λόγο. Με χαρά σας δίνω τον λόγο, κύριε Βίτ. Παρακαλώ. Χωρίς μικρόφωνο ο μιλητής, χωρίς μικρόφωνο. Μικρόφωνο. Χρησιμοποιήστε το μικρόφωνο παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Εξ ονόματος λοιπόν των περιφερειακών τμήματων ε, Θήρας Ανατολικής Σαξονίας Κέντρου Δράσης για τον ε, την επανεγκατάσταση λύκων στη Γερμανία σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση να εξεταστεί αναφορά μας. Για πρώτη φορά έχουμε τέτοια θέματα πολιτικής κυνηγίου και τονίζουμε ότι αυτά τα θέματα μπορούν να συζητούνται μόνο με τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων. Δυστυχώς δεν ε, ε τίνουν όλοι ευήκον ους σε τέτοιες, δράσει. δράσεις. Από τότε που υποβλήθηκε η αναφορά μας ε, πέρυσι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνεχίστηκε η ραδαία εξάπλωση των λύκων στη Γερμανία. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητα μια επιτυχία των οδηγιών για την προστασία των ειδών και της φύσης. Το τονίζω αυτό. Τονίζω επίση ότι θεωρούμε ακράδαντα, πιστεύουμε ακράδαντα ότι οι λύκοι όπω και τα άλλα αγρία ζώα έχουν δικαίωμα να ζουν σε αγέλε και ομάδε ώστε να μπορούν να επιβιώσουν και να συνεπάρχουν με του ανθρώπου στο φυσικό, φυσικό τους οικοσύστημα. Όμω η επιτυχία αυτή δημιουργεί και προβλήματα, σοβαρά προβλήματα, όπω γνωρίζουν πολύ καλά οι κτηνοτρόφοι που υφίστανται τι ε, αυξημένε απώλειε των ζώων του και μια απώλεια ποιότητα ζωή ε, που σημαίνει αυτό Επιπλέον, απώλεια ελαφιών, απώλεια επίσης ηθαγενών εγάγρων ή κρικρή, έστω αν θέλετε, μέσω των λύκων τα διαπιστώνουν όλα οι κυνηγοί. Ταυτόχρονα βέβαια υπό το πρίσμα της βιοπικιλότητας ακόμα και ο σημαντικός περιορισμός της προσωπικής ελευθερίας, σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη, ένα τρίτο των περιφερειών, των όσων ερωτήθηκαν από περιφέρειες που υπάρχουν λύκοι, εκφράζουν φόβους για να περπατούν στη φύση, καθώς επίσης και για την αύξηση του κινδύνου του λύκου για τους ανθρώπους. Και αυτό έχει μειώσει την αποδοχή των λύκων από πλευράς των πολιτών μας. Έτσι βλέπουμε λοιπόν ότι αυτό δεν είναι μια ε, σωστή μακροπρόθεμη στρατηγική για τους λύκους. Δικός μας στόχος είναι να αλλάξει η διαχείριση και με μια νέα διαχείριση να βελτιώσουμε την προσαρμογή και την αποδοχή σε σχέση με τους λύκους και τη φύση μέσα από μια στρατηγική προστασίας. Ένας άλλος ε, στόχος ε, σε σχέση με την, για την προστασία του λύκου δεν μπορεί να επιτευχθεί με διαφορετικό τρόπο. Είμαστε πισμένοι ότι μόνο μια ρύθμιση του, του αριθμού των λύκων μπορεί να δώσει λύσεις σύμφωνα με τις ε, διεθνείς ρυθμίσεις και κανονισμούς ένα πληθυσμό λύκων που σήμερα <clears throat> δεν δημιουργεί κινδύνους στην Ευρώπη. Όταν λάβουμε υπόψη 10.000 λύκους για παράδειγμα που ζουν ελεύθερα, ελεύθεροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σύμφωνα με το IUCN του 2004 που χαρακτηρίζει τους λύκους ως μη ε, ε, επαπειλούμενο είδος ε, πλέον. Σύμφωνα με τις ευνοϊκές αυτές συνθήκες για, τις φυσικές, για τη φυσική διαβίωση του λύκου και όσον αφορά και το 2013 και έρευνα που έγινε στην Πολωνία ή σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο Όρχους στη Δανία πέρυσι δείχνουν ότι αυτοί οι λύκοι που ζουν στην ε, Γερμανία και στη Δυτική Πολωνία καθώς επίσης και στην ε, ε, περιοχή της Βαλτικής μέσω της μετανάστευσής τους μπορούν να ανταλλάξουν το γενετικό τους υλικό και με αντικειμενικούς επιστημονικούς όρους ζητούμε να δείξετε κατανόηση εσείς ως Ευρωβουλευτές και να υποστηρίξετε εμάς ως τους αρμόδιους για τα θέματα θύρας. Συνοψίζοντας θέλω να πω με τη δική μας αναφορά εμείς οι κυνηγοί από την Ανατολική Σαξονία είμαστε υπέρ της μεταφοράς από το παράρτημα 4 της οδηγίας στο παράρτημα 5 ως έναν αναγκαίο όρο για μια σωστή απόφαση για τη βιοπικιλότητα. Θέλουμε να ληφθεί μια σωστή απόφαση για την κοινωνική βιωσιμότητα του λύκου. Ο λύκος μπορεί, ε, μια και είναι θηρευτής, ε, δεν μπορεί να είναι δεκτός ε, παντού και χωρίς όρους και προορισμούς. Όμως έχουν δικαίωμα να ζουν σε βιώσιμες αγέλες και ομάδες ηλίκη. Χρειάζεται ένα, ένας αριθμός πληθυσμού λύκων που διασυνοριακά θα μπορεί να επιβιώσει μέσω εποπτείας και παρακολούθησης όλα τα επιστημονικά αντικειμενικά στοιχεία για τον αριθμό του πληθυσμού των ε, λύκων πρέπει να παρακολουθηθούν. Είναι απαραίτητος και ένας διάλογος με τους εμπλεκόμενους ε, κυνηγού. Ε, εμείς εκφράζουμε την προθυμία μας ως θέμα αρχίσει για να έχουμε αυτή την ανταλλαγή απόψεων περιφερειακά, τοπικά και εθνικά για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στι σχέσει μεταξύ ανθρώπου και λύκου. Και φυσικά βρισκόμαστε, ευθυγραμμιζόμαστε με την, τις αποφάσεις που ελήφθησαν στη Δρέσδη με τα έγγραφα σε σχέση με το Positions Papier Wolf, δηλαδή τα έγγραφα εργασία για τον Λύκο. Ευχαριστώ. Thank you very much. I give the floor to the Commission. Ευχαριστώ πολύ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ξεκινήσω με, με ένα προκατακτικό σχόλιο γιατί και αυτοί και, και, αυτοί και οι επόμενες αναφορές δείχνουν ε, πόσο δύσκολο είναι σήμερα, δύσκολη είναι σήμερα η διατήρηση των μεγάλων κινηδών και συγκεκριμένα των λύκων. Από απόψεως νομοθετικής, τα μεγάλα σαρκοφάγα μεταξύ των οποίων και οι λύκη είναι τμήμα της ε, κληρονομιάς βιοπικιλότητας Ευρωπαϊκής Ένωσης και ένα ε, τμήμα της ε, ευρωπαϊκής ιστορίας για τον των οικοσυστημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι σημαντικός ο ρόλος του. Επειδή έγινε προσφάτως αποκατάσταση των μεγάλων αυτών σαρκοφάγων, δεν σημαίνει βέβαια ότι η πολιτική διατήρησή μας ήταν απολύτως επιτυχής. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωρίζει ότι αυτό το συγκεκριμένο είδος, συγκεκριμένα ηλίκη, ε, σε περιοχές από τις οποίες ε, έλειπαν τεράστιες, για τεράστιες περιόδους, όπως 100 χρόνια για παράδειγμα, στην Γερμανία, έχει ε, σχέση με κάποιες συγκρούσεις ε, που αφορούν για παράδειγμα ε, την απειλή στα παραγωγικά ζώα, ανταγωνισμός ή τέλος πάντων καζόμενος ανταγωνισμός με το κυνήγι, με διάφορα άλλα είδη και όπως επίσης και ε, ε, διάφορους φόβους ε, όπως συμβαίνει για παράδειγμα με τις αρκούδες. Είμαστε υποχρεωμένοι να το αναγνωρίσουμε και πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να ελαχιστοποιήσουμε όλες αυτές τις συγκρούσεις και να αυξήσουμε την αποδοχή των λύκων από το κοινό και να λάβουμε υπόψη βέβαια και τα ε, συμφέροντα των ε, πληθυσμών της ε, υπαίθρου. Ένα από τα ζητήματα αυτής της αναφοράς ήταν οι απώλειες σε παραγωγικά ζώα. Πρέπει να πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συστηματικά δεν λαμβάνει πληροφορίες σε σχέση με απώλειες παραγωγικών ζώων από τα κράτη-μέλη. Δεν υποχρεωμένα να παρέχουν τις πληροφορίες αυτές, όμως έχουμε κάποια στοιχεία από τη Γερμανία, γιατί πριν από μερικά χρόνια ζητήσαμε μία μελέτη από την Ευρωπαϊκή, από Ευρωπαίους για τα μεγάλα σαρκοφόγα, σαρκοφάγα και από τα δεδομένα αυτά που αφορούν τη Γερμανία βλέπουμε ότι οι απώλειες ε, παραγωγικών ζώων είναι χαμηλές για τη Γερμανία σε σχέση με άλλες γειτονικές χώρες. Τα αριθμητικά στοιχεία που έχουμε για το 2011 για παράδειγμα είναι περίπου 225 ε, παραγωγικά ζώα που αποτέλεσαν λία, ε, κυρίως πρόβατα, ε, από λία λύκων, κατέτος. Και γνωρίζουμε επίσης ότι στη Γερμανία τέτοιου είδους απώλειες είναι αντικείμενο αποζημίωσης από τις δημόσιες αρχές και γνωρίζουμε επίσης ότι στη Γερμανία ε, οι αρχές έχουν ε, δημιουργήσει ένα σύστημα για την προστασία και την πρόβλεψη, μέτρα πρόβλεψης και μιλάω για ηλεκτροφόρα σύρματα ε, ακριβώς για να μην είναι τα παραγωγικά ζώα λία των λύκων. Επίσης γνωρίζουμε ότι η Γερμανία και συγκεκριμένα, το συγκεκριμένο κρατήδιο χρησιμοποιεί ε, χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υποστήριξη τέτοιου είδους ε, προληπτικών μέτρων και αναφέρομαι στα προγράμματα ανάπτυξης της ε, Σαξονίας όπως επίσης και σύμφωνα ε, με τα δεδομένα που έχει λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τις γερμανικές αρχές, μιλάμε για μία, ε, ένα πολύ μικρό επαπειλούμενο πληθυσμό ο οποίος δεν βρίσκεται σε καθεστώς διατήρησης και σύμφωνα με την πρόσφατη εκτίμηση του καθεστώτος διατήρησης ε, για την περίοδο 2007 με 2012 μιλάμε για 39 ε, λύκους στη Γερμανία. 39 λύκους, ε, μια άλλη πηγή που λαμβάνει υπόψη στοιχεία 2011 ε, και 2012 αφορά 43 ενήλικες λύκους. Δεν έχουμε να κάνουμε με μεγάλο πληθυσμό, μιλάμε για μικρό πληθυσμό που βρίσκεται υπό απειλή. Και σύμφωνα με την οδηγία ε, περί οικοσυστημάτων ε, πρέπει να υπάρξει αυστηρό καθεστώς προστασίας, δηλαδή να απαγορεύεται το κυνήγι βάσει της οδηγίας περί οικοσυστημάτων. Όμως ένα κράτος μέλος μπορεί να ε, παρέχει εξαιρέσεις και σε αυτή την περίπτωση υπό συγκεκριμένες συνθήκες που προβλέπει η οδηγία και δεδομένου βέβαια ότι αυτό δεν υπονομεύει την επίτευξη ενός ε, ε, ε, μιας διατήρησης του πληθυσμού στην φυσική του διανομή. Όσον αφορά τώρα την αλλαγή της νομοθεσίας και την αλλαγή του νομικού καθεστώτος του λύκου στη Γερμανία, που σύμφωνα με τον αναφέροντα θα έπρεπε να περάσει από το να, να, να περάσει από το παράρτημα 4 στο παράρτημα 5 που θα επέτρεπε τη διαχείριση, δηλαδή το κυνήγι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν συμμερίζεται την άποψη αυτή για τους λόγους που εξηγήσαμε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν προγραμματίζει τροποποίηση των παραρτημάτων ε, της οδηγίας περί οικοσυστημάτων. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ... Ε, σας ευχαριστούμε πολύ. Αρχίζουν οι παρεμβάσεις των Ευρωβουλευτών. Βαλέρο παρακαλώ. Σα ευχαριστώ πολύ. Πολύ χαίρομαι, Πρόεδρε, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ότι δεν στοχεύει να αλλάξει την οδηγία. Εγώ κατοικώ σε μια περιοχή στη Σουηδία όπου υπάρχουν αρκούδες και λύκοι σε μεγαλύτερο βαθμό, σε μεγαλύτερο ποσοστό από στην υπόλοιπη Σουηδία. Το κυνήγι των αρκούδων και λύκων είναι κάτι το πολύ ζωντανό σε εμάς. Ε, με ιδιαίτερο ιδιαίτερος αριθμός πολιτών ασχολείται με αυτό. Μια τώρα άλλη οδηγία δεν χρειάζεται τροποποίηση οδηγίας. Ε. Η συζήτηση στοχεύει στο ότι αυτοί οι πληθυσμοί ζώων πρέπει να προστατεύονται. Πολλοί άνθρωποι βέβαια φοβούνται τους λύκους ε, και δεν έχουν συνηθίσει να υπάρχουν λύκοι γύρω τους στη φύση. Γίνεται επίσης όμως και λόγος για την προστασία της φύσης ε, και των ε, ζώων των κτηνοτρόφων. Έχουμε όμως μεθόδους όπως οι ηλεκτρικούς φράχτες, ε, ηλεκτροσύρματα που ηλεκτροδοτούνται για να προστατεύονται αυτά τα ζώα. Ουσιαστικά έχουμε μια κατάσταση που παλιότερα δεν υπήρχε. Και στη δική μου περίπτωση, εκεί δηλαδή όπου κατοικώ εγώ στη Σουηδία, ο λύκος μπορώ να πω ότι είναι ένα επιπλέον ζώο όπως ο τάραδος για παράδειγμα που ε, ε, κυνηγά ας πούμε τον τάραδο. Υπάρχει μια ας το πω έτσι ανταγωνιστική σχέση και αυτό είναι και ίσως ένα αίτιο για προβλήματα που υφίστανται. Δεν μπορούμε να πούμε ότι εμείς οι ίδιοι θέλουμε να κυνηγούμε και τελεία και παύλα γι' αυτό χρειάζεται κάποια ρύθμιση. Υπάρχουν κάποιοι που είναι κυνηγοί, σίγουρα. Όμως πρέπει από την άλλη πλευρά να είμαστε και πρόθυμοι να λάβουμε υπόψη και την ε, ύπαρξη άλλων ε, ζώων, όχι μόνο των ταράνδων, αλλά και των λύκων στην ε, περιοχή μας. Και πρόσφατα, κατά την τελευταία περίοδο, συνέβη το εξή. ότι προτιμούσαν να προστατεύεται ο τάραδο οι πολίτε, αλλά όχι ο λύκο. Αν όμω θέλουμε να προστατεύεται ο τάραδος πρέπει να προστατεύεται και ο λύκο. Αυτό πιστεύουμε εμεί δεν υπάρχει, ας το πω έτσι, κάποιο, μ, κάποιος πληθυσμός λύκων που θα μπορούσε να δικαιολογήσει μια τροποποίηση της οδηγίας. Βαλένσα παρακαλώ. Λάθος έκανα, εσείς έχετε τον λόγο παρακαλώ. Ε, yeah, Σε ε, ε, ευχαριστώ και εγώ πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα θερμά να ευχαριστήσω για τους συντάκτες αυτών των αναφορών, για το ότι κατέθεσαν αυτές τις αναφορές σε μας. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να, να επιστήσουν την προσοχή μας στην κατάσταση των λύκων και είναι και καλό το ότι έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη το ζήτημα των λύκων. Είναι σημαντικό αυτό γιατί, διότι ο λύκος αποτελεί συστατικό στοιχείο της φύσης μας και ανήκει στη φύση αυτή όμως οι λύκοι απειλούνται ιδιαίτερα όσον αφορά την ίδια την επιβίωσή τους. Από πολλές περιοχές και περιφέρειες έχουν εξαφανιστεί, εξαφανίζονται. Τους κυνηγούν ανελαίητα οι άνθρωποι και τους εξοντώνουν. Είναι ουσιαστικά ένα, ένα θαύμα θαύμα μπορεί να το αποκαλέσει κανείς ότι δεν ε, ε, εκριζώθηκαν, δεν εξοντώθηκαν τελειωτικά οι λύκοι στην Ευρώπη. Μπορούμε να εκφράσουμε την ικανοποίησή μας λοιπόν ότι εξαπλώνονται οι λύκοι στην ε, Ευρώπη σήμερα και μπορούν να επιβιώσουν και πρέπει να θεωρήσουμε ότι αυτό μας, πρέπει να μας κάνει να εκφράζουμε την ικανοποίησή μας. Όχι μόνο όσον αφορά την κατάσταση στην Σουηδία, Γερμανία ή και αλλού, αλλά επίσης και σε χώρες όπου οι λύκοι εδώ και δεκαετίες δεν είχαν ξαναπαρουσιαστεί. Εντάξει, ωραία, στην Ολλανδία είναι όλα σχεδόν έχουν γίνει, ε, είναι, είναι πόληση μια πίσω από την άλλη, αστικά κέντρα. Ωστόσο, εκεί κοντά όπου ζω εγώ, είδαν κάποιοι έναν λύκο και η αντιμετώπιση των πολιτών δεν ήταν ε, τόσο επιθετική. Δεν ήταν, οι, οι λιγότεροι διαρωτήθηκαν γιατί να υπάρχει εδώ ένας λύκος. Κανεί δεν είπε ότι οι λύκοι θα επιτίθεντο κατά ανθρώπων και άρα λοιπόν είναι γι' αυτό και μόνο τον λόγο επικίνδυνοι. Δεν είναι επικίνδυνοι οι λύκοι αφεαυτών, δεν τρώνε μικρά κορίτσια ή δεν κινδυνεύουν γιαγιαδε από αυτού. Αυτά τα παραμύθια πρέπει να πάψουν να υπάρχουν, να διαδίδονται πλέον. Φυσικά ωραία, τρώνε κάποια ζώα, πρόβατα, καθήκια, κουνέλια, λαγού ε, οι λύκοι. Πολύ καλά. Μπορούν επίσης ε, και ε, αγελάδες ε, βόδια να, να επιτεθούν εναντίον τους και να τα κατασπαράξουν. Έχουν την ευθύνη τους όμως οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι να προστατεύουν τα ζώα τους. Όπως έχουν και ευθύνες να προστατεύουν και τους φυσικούς, την φύση γύρω τους. Και εμείς έχουμε ως πολιτικοί τις ευθύνες μας. Πρέπει και εμείς να μεριμνήσουμε να γίνει μια έρευνα που να είναι αποτελεσματική όσον αφορά τον πληθυσμό, τους πληθυσμούς των ε, ε, ζώων αυτών. Να μην βασιστούμε μόνο στα στοιχεία που μας ε, δίνουν οι κυνηγοί χρειάζονται αντικειμενικές επιστημονικές μέθοδοι παρακολούθησης και αξιολόγησης και εποπτείας φυσικά και παρακολούθησης. Χρειάζονται και κονδύλια, ένας προϋπολογισμός για την έρευνα για αυτές τις δράσεις, κονδύλια που θα διασφαλιστούν και θα διατεθούν. Πολλά ενδιαφέροντα πράγματα βρίσκονται καθοδόν και βρίσκονται υπό ανάπτυξη και εξέλιξη. Και αυτό όσον αφορά μελέτες, επίσης υπάρχει και η ευθύνη για να είναι βιώσιμη η κατάσταση της φύσης, να υπάρχει η αηφορία η φυσική και να υπάρχουν προοπτικές για τα άγρια ζώα όπως τους λύκους. Γι' αυτό δεν πρέπει να αποδυναμωθεί η οδηγία των βιοτόπων habitat οδηγία και από το αντίθετο πρέπει να συμβεί, να ενδυναμωθεί, να ε, ε, ενισχυθεί. Έχουμε ευθύνε όσον αφορά και την ε, διαφώτιση των πολιτών, πληροφόρηση και ενημέρωσή τους. Ας μην αρχίσει να ισχύει εδώ το παραμύθι της κοκκινοσκουφίτσας για τους λύκους. Ας αφήσουμε λοιπόν τα των λύκων των λύκων. Ε, και δεν θα χρειάζονται λοιπόν τότε και οι κυνηγοί να σκοτώνουν όλα αυτά σε εισαγωγικά τα επικίνδυνα ζώα. Κυρία Πρόεδρε, λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο θα ήθελα να ολοκληρώσω και να πω ότι με σαφήνεια υπήρξε η τοποθέτηση. Δεν έχουμε κάποια πρόθεση να αλλάξει η κατάσταση όσον αφορά τους λύκους. Αδημονώ να δω το τι θα γίνει για να μπορέσει να ενδυναμωθεί η παρουσία των λύκων και ο πληθυσμός τους. Σας ευχαριστώ. Νομίζω συμφωνούμε όλοι πρόεδρε ότι είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα αυτό και δεν θέλουμε να εξοντώσουμε τους λύκους όπως είχε συμβεί στο παρελθόν. Όμως πρέπει να λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι αυξάνεται ο πληθυσμός των λύκων σήμερα και αυτό έχει τις επιπτώσεις του ως γεγονός όσον αφορά τον αριθμό άλλων ζώων στην φύση. Και γι' αυτά για όλα αυτά η Επιτροπή νομίζω διεξοδικά παρουσίασε τα θέματα, αλλά ακόμα και εκεί άκουσα ότι δεν υπάρχουν λέει αρκετά επιστημονικά στοιχεία για να μας δώσουν μια βάση ε, ε, που να είναι επαρκής από πλευράς πληροφοριών και επιστημονικά. Τούτων λεχθέντων, συμφωνώ με την συνάδελφο, χρειαζόμαστε περισσότερη έρευνα, περισσότερες πληροφορίες. Καλή ιδέα θα ήταν άμεσα να απευθυνθούμε και να ε, ρωτήσουμε εμείς, ε, να ζητήσουμε εμείς ως Κοινοβουλευτική Επιτροπή από τις αρμόδιες αρχές, ίσως τους αρμόδιους, τον αρμόδιο Υπουργό στη Γερμανία, να θέσουμε συγκεκριμένες ερωτήσεις για τον αριθμό των ζώων, για παράδειγμα για το τι συμβαίνει με την, τις επαφές ε, λύκων Γερμανία, στη Γερμανία με λύκους της Πολωνίας και όλα αυτά θα είναι δυνατόν να απαντηθούν με ερωτήσεις που θα διατυπώσουμε για να δημιουργήσουμε τη μεγαλύτερη εικόνα, να κατανοήσουμε συνολικά την κατάσταση αυτών των ζώων, των λύκων. Διότι πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι ήταν απειλούμενο είδος η λύκη κατά το παρελθόν. Και γι' αυτό ακριβώς είναι ένα είδος που έχει κάθε λόγο να ε, μπορέσει να επιβιώσει και μπορεί να θεωρηθεί αξιόλογη επιτυχία η επιβίωσή του. Θα πρέπει να δούμε πόσο ο αριθμός αυτών των ζώων που αυξάνεται μπορεί να αντιμετωπιστεί με τον καλύτερο τρόπο για μας τους ανθρώπους και για το περιβάλλον, για τη φύση. Περισσότερες πληροφορίες λοιπόν χρειαζόμαστε θα έλεγα. Ευχαριστώ. Okay, um... Πρόεδρο σας ευχαριστώ. Λοιπόν όλοι φαίνεται. Θα πρέπει τώρα να δώσω το λόγο στον αναφερόμενο πάλι και μετά να προσπαθήσουμε να κλείσουμε το θέμα. Οι συνάδελφοι δεν βοήθησαν ιδιαίτερα. Θα δώσω το λόγο στον αναφερόμενο τώρα. Χωρίς μικρόφωνο, χωρίς μικρόφωνο. Yeah. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα να πω δύο λόγια. Καταρχήν ευχαριστώ γιατί μπόρεσε να εξεταστεί αυτό το θέμα στο Ευρωκοινοβούλιο. Εντυπωσιάστηκα και για την απήχηση την οποία βρήκε αυτό το θέμα. Όχι όμως ε, δεν συμφωνώ επί του θέματος με κάποιες τοποθετήσεις που έγιναν όμως. Από τον πρώτο που παρενέβη που επειδή ε, δεν μπόρεσα να καταλάβω πλήρως ε, α, τα όσα είπε αν τοποθετούμενος για τους αριθμούς των λύκων στη Γερμανία λέγεται κάτι, τότε πρέπει οι σωστοί αριθμοί να αναφέρονται. Οι σωστοί αριθμοί του γραφείου Λύκου, Λούπους στη Γερμανία, που είναι υπεύθυνο στη Σαξονία για την παρακολούθηση, την εποπτεία, λέει ότι το 2013 31 γέλες υπήρχαν και ζούσαν στη Γερμανία. 31 γέλες και 12 από αυτές στη Σαξονία. Η Σαξονία λοιπόν είναι η πολυαριθμότερη πολιτεία, το πολυαριθμότερο κρατήριο όσον αφορά τον αριθμό των ε, λύκων. 31 αγέλες. Τουλάχιστον 5 ή και 10 ζώα μπορεί να έχει μια αγέλη. Υπολογίστε αριθμητικά πόσα είναι λοιπόν με 31 αγέλες, με 10 η κάθε αγέλη. Από την άλλη μεριά τώρα, το αν επαπειλείται ένα είδος ή όχι από γεωγραφικούς λόγους δεν πρέπει να κρίνουμε μόνο με γεωγραφικά επιχειρήματα. Πρέπει σε σχέση με τον ίδιο τον πληθυσμό των ζώων να, κάνουμε, να βγάζουμε τα συμπεράσματά μας. Και έτσι και ως υπεύθυνοι για τη φύση να αναφέρουμε τον αριθμό αυτών του πληθυσμού των ζώων σε σχέση με τη φύση στην οποία ζει για να δούμε αν υπάρχει συμβατότητα ή όχι και συνάδει ο αριθμός με τη φύση διότι εδώ βρίσκονται σε μια αντιστοιχία ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος, να μην επαπειλείται ούτε η φύση ούτε ο λύκος. Και θα πρέπει να περάσει η εντύπωση από ό,τι φαίνεται στο Ευρωκοινοβούλιο ότι υπό το πρίσμα κατοίκων των πόλεων οι πληθυσμοί της υπαίθρου δεν μπορούν να γίνουν, να, να αντιληφθούν οι κάτοικοι των πόλεων αν τα θεμητά τους αυτά αιτήματα για το αν είναι επικίνδυνος ο λύκος ή όχι, αν τοποθετούμεθα με αυτόν τον τρόπο όπως ακούστηκε και θεωρείται ότι είναι αυλαβές ζώο ο λύκος, ε, δεν ισχύει αυτό. Δεν κυνηγά τον άνθρωπο ο λύκος σίγουρα. Γνωρίζουμε όμως ότι είναι σε θέση να σκοτώσει άνθρωπο ο λύκος όταν αναγκαστεί και υπάρχουν τεκμηριωμένες περιπτώσεις θανάτων από, ανθρω... λύκους των ανθρώπων και ήταν 69 επιθέσεις συνολικά και που πολλές φορές ήταν θανάσιμες οι επιθέσεις αυτές. Αν κάποιος λοιπόν ισχυριστεί έτσι ότι λέει, λέει η γιαγιά ότι υπέστη κάποια επίθεση ο άνθρωπος από τον Λύκο και αυτό δεν ισχύει σήμερα και είναι παροχημένο δεν μπορεί να ισχύει αυτό συλλήδιν έτσι και είμαστε υπέρ του ότι η ανταλλαγή πληροφοριών που ξεκίνησε με αυτόν τον τρόπο πρέπει να βελτιωθεί σημαντικά με συμπερίληψη όλων εκείνων που ζουν στις περιοχές της υπαίθρου και θέλουν να ζουν από κοινού και να συμβιώνουν με τους λύκους, ιδιαίτερα δηλαδή τους κα, κατοίκους της υπαίθρου. Ευχαριστώ. Thank you for having... Ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστούμε που συμμεριστήκατε τα βιώματά σας μαζί μας. Αν θυμάμαι τα παιδικά μου χρόνια στην Σουηδία και του συγγενείς μου που το φθινόπωρο έβγαιναν για κυνήγι, τουλάχιστον μπορούμε να πούμε ότι στη χώρα μου υπάρχουν πολλά περισσότερα θύματα και ζημιά, ζημιές που προκαλούνται από τις αρκούδες, πολύ περισσότερες από ό,τι από τους λύκους. Την άλλη φορά μπορεί να έχουμε μία αναφορά για τις αρκούδες, ποιος ξέρει. Ίσως λοιπόν όμως είναι πιο δύσκολη η προσέγγιση αυτή του, της επικίνδυνης αρκούδας επειδή όλοι γνωρίζουμε το αρκουδάκι το οποίο έχουν στην αγκαλιά τους τα παιδιά και τα μωρά. Λοιπόν, παρόλα αυτά, εν πάση περιπτώσει, θα ήθελα να προτείνω δεδομένου ότι είναι μια πρόκληση αυτό το θέμα και συγκινησιακά φορτισμένο, συναισθηματικά φορτισμένο θα μπορούσαμε να απευθυνθούμε στις αρχές της Σαξονία με μια επιστολή και να ζητήσουμε να υπάρξει να διάθεση επικαιροποιημένων στοιχείων που θα μας διατεθούν για όλα τα στοιχεία και τους αριθμούς, αριθμητικά μεγέθη για την κατάσταση των λύκων. Και θα παρακολουθήσουμε επίσης το τι συμβαίνει σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ποια συνέχεια δίνεται. Θα θέλαμε να ξέρουμε αν θα πρόκειται να υπάρξει κάποια γραπτή τέτοια ε, κοινοποίηση σε εμά πληροφόρηση ή όχι. Υπάρχει κάτι που θα θέλατε να μας πείτε από την Επιτροπή, παρακαλώ. Uh, yes, we might provide an... Ίσως να μπορέσουμε κάποια συμπληρωματικά στοιχεία να δώσουμε, να διευκρινίσουμε κάποια από τα θέματα, <coughs> αλλά αυτή τη στιγμή θα αναφερθώ σε κάποια από τα σημεία τα οποία τέθηκαν από τους αναφερομένους και τα οποία δεν σχολίασα προηγουμένως. Ο ανταγωνισμός ανάμεσα στους λύκους από τη μία και τους κυνηγού από την άλλη. Υπάρχει μια διάκριση το να γίνονται τα οικόσιτα ή παραγωγικά ζώα λία των λύκων, κάτι το οποίο θα έπρεπε να αποθαρρύνεται και να προβλέπεται και το κατά πόσο άγρια ζώα είναι λία των λύκων και αυτό είναι μια φυσιολογική διαδικασία την οποία δεν πρέπει να προβλέπουμε ούτε να αποθαρρύνουμε γιατί είναι τμήμα της λειτουργίας του οικοσυστήματος. Πάρα πολλοί κυνηγοί δεν συμφωνούν. Δεν τους αρέσει. Θεωρούν ότι υπάρχει ένας ανταγωνισμός ε, ειδικότερα από τους ε, λύκους. Όμως σήμερα στην Ευρώπη οι πληθυσμοί των ε, αγριόχειρων, των ταράνδων ε, έχουν αυξηθεί και συνεχίζουν να αυξάνονται. Είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι 50-100 χρόνια πριν. Επομένως η δική μας γραμμή είναι η εξής, ότι υπάρχουν πάρα πολλά είδη τα οποία μπορούν να κυνηγήσουν οι κυνηγοί και πάρα πολλά ζώα που θα μπορούσαν να είναι λία με επιτρεπτό τρόπο για τους λύκους. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να λαμβάνεται υπόψη όταν ε, ε, δίδονται οι άδειε για κυνήγι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είδατε αν ρωτάτε πάντοτε μπορεί να πάρετε απάντηση. Έτσι γνωρίζουμε ότι μπορεί ενδεχομένως να υπάρξει μια ανακοίνωση με περισσότερες και λεπτομερέστερες πληροφορίες. Σας ευχαριστούμε λοιπόν πολύ. Το σημειώνουμε, οπότε παραμένει ανοιχτή η αναφορά ε, εν ώψη νέων πληροφοριών και θα αποστείλουμε και αυτήν ε, την ε, επιστολή που θα ζητά περισσότερες πληροφορίες και αριθμητικά στοιχεία από τις αξονικές αρχές. Ούτως λοιπόν θα πράξουμε. Περνάμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά τον Ιβηρικό λύκο. Και θα ήθελα να μάθω ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στο Σκανδιναβικό και τον Ιβηρικό λύκο. Καταρχάς, μοιάζουν. Αναφορά υπαριθμών 1771 του 2013 εξ ονόματος του Λόμπο Μάρλι σχετικά με την οδηγία για τους οικοτόπους ε, και την προστασία του ιβερικού Λύκου και 2032 του 2013 για την παραβίαση της νομοθεσίας της Ένωσης για την προστασία των λύκων στην περιοχή Αστουρίας της Ισπανίας. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον Μαουρίθιο Αντών Ορτούζαρ. Έχετε το λόγο. Όχι πάνω από πέντε λεπτά παρακαλώ. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα, καλό σας βράδυ έστω. Να δούμε το βίντεο για να δείτε περί τίνος πρόκειται. Αυτά είναι τα βουνά στην Ισπανία. Είναι εκεί όπου βρίσκεται η πανίδα μας. And those are our wild Iberian wolves. Just imagine you are a nature lover from any country in Europe. You have... Αυτό σημαντικό για όλους όσους αγαπούν τη φύση. Έρχεται κάποιος στην Ισπανία να δει έναν τέτοιο λύκο, ιβυρικό λύκο και βλέπει μια ολόκληρη οικογένεια να παίζει στο λιβάρι, στο γρασίδι. Και μετά όμως βλέπει κανείς ότι μετά ε, πεθαίνουν μπροστά στα μάτια σας μετά με, με πόνους και αγωνία δύο λύκοι. Αυτό δεν είναι κάποιο παραμύθι. Έγινε κάποιες εβδομάδες πριν και δείχνει στον κόσμο στην Ισπανία το τι συμβαίνει. Ένα θέμα είναι το μέλλον, όπου διαδραματίζει το ρόλο του ο στους βιοτόπους, στη φύση και δημιουργεί και όρους προόδου με την, ε, το, την υπεύθυνη, ε, τις υπεύθυνες βιοκαλλιέργειες ε, και την καλλιέργεια του βιοτόπου. Το άλλο είναι το παρελθόν όπου έχουμε τους κυνηγού ε, και τους μανιώδεις κυνηγού με καιροσκόπους πολιτικούς που θέλουν να κερδίσουν ψήφους που διαδίδουν το μίσος κατά του λύκου μεταξύ των κτηνοτρόφων για να ε, ζήσει, επιζήσει ε, αιώνια ο μύθος του επικίνδυνου ζώου του λύκου και να αισθάνονται ε, οι υπόλοιποι. Είδατε λοιπόν τα, ε, ε, τα τελευταία ε, στοιχεία του David Attenborough για την εκπομπή του The Hunt όσον αφορά το κυνήγι και την οικολογία των, αυτών των θηρευτικών ειδών όπως παρουσιάστηκαν στα επεισόδια αυτά τα τηλεοπτικά. Έχουμε, πραγματικά θαυμάζουμε τα ζώα αυτά τα οποία είναι θηρευτές στην Αφρική και αλλού και πραγματικά βλέπουμε πόσα ε, τα ζώα της αγέλης μεταδίδουν στα νεότερα ζώα τις γνώσεις τους ώστε να μπορούν να κυνηγούν και εκείνα αποτελεσματικά καθώς ενηλικιώνονται. Φανταστείτε τις αντιδράσεις εκατομμυρίων θεατών αν θα μπορούσαν μετά από αυτές τις εκπομπές του Άτενμπορο να έβλεπαν τα, αυτά τα στιγμιότυπα από την Ισπανία με τον, ε, με τον θάνατο αυτό, επίπονο θάνατο των λύκων χωρίς να υπάρχει κανένας επιστημονικός λόγος θάνατοι που προκαλούν από αξιωματούχους του δημοσίου που τυχαία επιλέγουν κάποια ζώα να θανατώσουν ή από κυνηγούς που θέλουν ε, να θεωρηθούν ε, ε, πεπειραμένοι κυνηγοί και κυνηγούν και σκοτώνουν αυτά τα ζώα ώστε αντί να ε, είναι οι αποτελεσματικοί θηρευτές για τη διασφάλιση της ε, πανίδας να έχουμε μια ομάδα από προσανατολισμένων ζώων που επιτίθενται πολλές φορές ε, κατά των προβάτων και των ζώων των κτηνοτρόφων. Θα ζούσε κανείς έτσι ένα ταξίδι στον χρόνο από τον 21ο αιώνα προς τα πίσω προς μια αρχαΐζουσα ας το πω έτσι κατάσταση που θυμίζει τον 19ο αιώνα. Ο Ιβυρικός λίκος προστατεύεται ήδη στην Πορτογαλία, αλλά μας εκκλείσει δυσάρεστα ότι οι Πορτογαλικοί αυτοί λύκοι σκοτώνονται, σκοτώνονται, θανατώνονται όταν περνάνε τα σύνορα της Πορτογαλίας και εισέρχονται στην Ισπανία. Για να σταματήσει αυτό υπήρξε μια αναφορά ώστε να προστατεύσει το Ευρωκοινοβούλιο την προστασία του λύκου να την προωθήσει στο σύνολο της Ιβηρικής Χερσονήσου. Αν, θεωρείτε, αν δείτε τα στοιχεία της Ισπανικής κυβέρνησης θα πιστέψετε ίσως ότι ο λύκος ευτυχεί στην Ισπανία. Δυστυχώς δεν συμβαίνει αυτό. Εδώ έχουμε κάποια στοιχεία σχετικά. Πρώτον, το είδος δεν βρίσκεται σε ευνοϊκή κατάσταση διατήρησης ή συντήρησης. Σύμφωνα με το ίδιο το άρθρο 1 της οδηγίας για τους βιοτόπους, ευνοϊκές συνθήκες και όροι σημαίνουν να μπορεί το είδος να αυτοπροστατεύεται και να επιβιώνει ως άρρηκτα μέρος του βιοτόπου του. Όμως με το κυνήγι και τα λοιπά υφίσταται στρεβλώσεις η ολίκο σήμερα και δεν μπορεί να υλοποιήσει το ρόλο του. Η αυστηρή προστασία, απόλυτη προστασία είναι απόλυτα αναγκαία. Η εκτίμηση των, της κυβέρνησης για τους αριθμούς ε, των λύκων, η υπερβαίνει κατά 40 ή 50% τον πραγματικό αριθμό των λύκων. Μια, ένας τέτοιος υπερπληθωρισμός του αριθμού των λύκων είναι κίνδυνος ε, ως στοιχείο. Όταν βλέπουμε ότι υπήρξε μια στενοπός ε, ε, ε, μερικές δεκαετίες πριν και ότι αυτή η κατάσταση ε, διακυβεύει την δυνατότητα επιβίωσης ε, των άγριων αυτών ζώων, των λύκων, πρέπει να σταματήσει το αλόγιστο κυνήγι, ώστε να μπορέσουν να επιζήσουν οι λύκοι και να ανταλλάξουν το γενετικό του υλικό και να ευημερήσουν. Πρέπει να σταματήσει η σφαγή και να δώσουμε μια ευκαιρία στο μέλλον, να μην απογοητεύσουμε απογοητεύσουμε αυτή την ελπίδα λοιπόν. Ευχαριστώ. ευχαριστώ που μας είπατε, την, παρουσιάσατε την υπόθεση αυτή και μας δείξατε και εξαιρετικώς ε, εικόνες, εξαιρετικά τοπία. Είναι καλό να βλέπει κανείς το ότι υπάρχει. Η δεύτερη είναι της κυρίας Ροντρίγες. Έχετε το λόγο κυρία Ροντρίγες. Σας ευχαριστώ πολύ. Είμαι παρούσα επειδή η αναφερομένη, εγώ εμφαίνομαι ως αναφερομένη, αλλά η αναφερομένη ε, που ε, δεν ε, παρίσταται και επιπλέον για την κατάθεση αυτής της αναφοράς του 2013 είχαμε τεχνική υποστήριξη αρκετών φορέων και ενώσεων περιβαλλοντικών στην Ισπανία και υποστηριχθήκαμε από χιλιάδες υπογραφές ε, υπέρ της, ε, ε, του αιτήματό μας. Στη δική μας αναφορά καταγγέλουμε την παραβίαση παρατυπιών που δείχνουν ότι υπάρχει παραβίαση κοινοτικού δικαίου. Πρώτον, παραβίαση όσον αφορά την διάθεση, τη δημοσιοποίηση των στοιχείων που δίνουν άδεια στην θανάτωση των λύκων. Και έτσι λοιπόν παραβιάζεται η δημοσιοποίηση και ε, γνωστοποίηση αυτών των στοιχείων. Δεν δημοσιεύονται τα στοιχεία αυτά στις ανακοινώσεις και στις ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρονται κάποιες από αυτές όσον αφορά το εθνικό, τον εθνικό δρυμό των κορυφών των Πυρηναίων, πίκος στην όμως ε, εδώ πρέπει να δούμε ότι πρόκειται για άλλο θέμα. Δεν δημοσιεύονται λοιπόν οι αποφάσεις ε, που δίνουν την άδεια να θανατώνονται γενικά οι ηλίκοι στην ε, περιοχή των Αστουριών. Πρόσφατα, χάρη στην δράση πολιτικών κομμάτων στο Κοινοβούλιο των Αστουριών και επειδή νέοι βουλευτές ε, που εισήλθαν σε αυτό το κοινοβούλιο ζήτησαν να υπάρξει η γνωστοποίηση αυτών των στοιχείων, επιτέλους μετά από πολλά έτη, μια και που ζητούσαμε αυτή την γνωστοποίηση, υπήρξε η αποκάλυψη αυτών των στοιχείων που αποδεικνύουν αυτό το οποίο εμείς καταγγέλουμε και καταγγείλαμε εδώ για τη θανάτωση των δίκων. Η δεύτερη παραβίαση είναι η μη σύνταξη έκθεσης αναδιετία όπως ε, ε, απαιτείται και δεν τηρείται η διάταξη του αντίστοιχου άρθρου. Οι Αστούριες δεν υλοποιούν αναδιετία αυτές τις εκθέσεις και έτσι δεν υπήρχε δυνατότητα από πλευράς του ε, Υπουργείου να υπάρξει κάποια ας το πω έτσι αναφορά σε αυτά τα στοιχεία μια και δεν διαβιβάστηκαν και δεν υπάρχει αντίδραση σε αυτή την παρατυπία την οποία αναφέρουμε από πλευρά της Επιτροπής. Και στα έγγραφα 4 και 5 α, σημειώνουμε δημόσια έγγραφα στα οποία η ίδια η υπεύθυνη αναγνωρίζει ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για τα, τη θανάτωση, τη θανατώση των λύκων και πληροφορίες ε, διαθέσιμες ε, για τα αίτια των ε, θανάτων. Είναι πολύ δύσκολο λοιπόν να υπάρξει μια εκπόνηση εκθέσεων με τέτοιου είδους απουσία στοιχείων. Το τρίτο στοιχείο το οποίο καταγγέλουμε είναι ότι μέσα στη ζώνη φυσικής διάδοσης δεν υπάρχουν ε, τα αντίστοιχα στοιχεία. Όσον αφορά και πριν από το 2002 και φέτος το 2015 ακολουθούνται πολιτικές που περιορίζουν τους λύκους ε, σε περιοχές ε, που βρίσκονται κοντά στο δίκτυο Natura 2000 φύση 2000 και στα υπόλοιπα, στα πράσινα ε, ως ζώνες, ε, τα υπόλοιπα που είναι σε λευκό ζώνες, είναι εκείνα τα οποία θεωρούν ζώνες ελεύθερες ε, από τους λύκους και έχουν εκεί σε σχέση με τους πληθυσμούς λύκων δεν υπάρχουν εκεί ε, λύκοι. Υπάρχει λοιπόν σαφής παραβίαση του κοινοτικού δικαίου δεν λέμε ότι δεν χρησιμοποιούνται μη επιλεκτικές μέθοδοι. Λέμε ότι γίνεται αδιάκριτη χρήση από πλευρά ε, των κρατικών αρχών για ειδικών δράσεων για την εξόντωση όλων των λύκων στις λευκές ζώνες που εμφανίζονται εδώ ως λευκές ζώνες διότι βλέπουμε ότι στο ε, δίκτυο ε, φύση 2000 ε, είναι ζώνες που είναι δύσκολη η διατήρηση, η συντήρηση τέτοιων πληθυσμών. Επίσης παραβίαση της υποχρέωσης να αναφέρεται ότι η έλεγχη πληθυσμών είναι η μόνη και ικανοποιητική λύση για να αντιμετωπιστούν οι ζημιές, οι απώλειες στο κεφάλαιο το κτηνοτροφικό των κτηνοτρόφων. Αυτό παραβιάζει το αντίστοιχο άρθρο της οδηγίας για τους βιοτόπους, για τα habitats. Θέλουμε να ξέρουμε πώς είναι δυνατόν σε σχέση με τις ε, αρχές της Αστούριες ε, να γίνει αυτό αξιόπιστο, μια και δεν υπάρχουν άλλα μέτρα τα οποία να λαμβάνονται. Δεν είναι λοιπόν η αδιάκριτη θανάτωση λύκων η μόνη λύση. Αυτό το οποίο εμείς ε, έχουμε ως απόδειξη, ως τεκμήριο υπαριθμών 10, αναφέρει ότι το κύριο συμπέρασμα και έχει αποδειχθεί αυτό επιστημονικά είναι ότι όσο περισσότερες θανατώσεις υπάρχουν τόσο μεγαλύτερες ζημιές γίνονται στο ζωικό κεφάλαιο των κτηνοτρόφων. Διότι αποδομούνται οι αγέλες κοινωνικά και εμφανίζονται μονασικοί λύκοι, οι οποίοι τρέφονται ακριβώς από τέτοιου είδους ε, ζώα όπως τα πρόβατα, οι αγελάδες, το ζωικό κεφάλαιο των κτηνοτρόφων που σκοτώνουν. Πρέπει λοιπόν εδώ να δούμε σε σχέση με τις περιβαλλοντικές πτυχές πρέπει να ανοίξει μια τέτοια προσφυγή ακριβώς εις βάρος της Ισπανίας και πρέπει να εξηγιανθεί αυτή η κατάσταση και εκφράζουμε την ικανοποίησή μας γι' αυτό. Επίσης εκφράζουμε τη βαθύτατη θλίψη μας για αυτές τις πολιτικές εξόντωσης των λύκων στις Αστούριες σε αυτή την περιοχή δεν γίνεται χρήση των, δημόσιων, των χρημάτων των φορολογουμένων για να χρηματοδοτηθεί κάποιο πρόγραμμα για την ειρηνική συμβίωση ζώων και ανθρώπων και παρόλα αυτά δίνονται τεράστια κονδύλια, ένα εκατομμύριο ευρώ για να μ, πληρώνονται αποζημιώσεις ε, για τις απώλειες, υποτιθέμενες αυτές απώλειες ε, των, ε, του ζωικού κεφαλαίου να, μην, να αναφέρω ότι δεν υπάρχει ούτε ένα κέντρο αποκατάστασης ε, όσον αφορά την πανίδα για παράδειγμα και για παράδειγμα για την αποστολή ζώων σε μικρές κλινικές. Αυτή είναι η κατάσταση όσον αφορά την πανίδα στην περιοχή μας. Θα ήθελα να ολοκληρώσω λέγοντάς σας κάτι ότι έχουμε πολλαπλά στοιχεία τα οποία έχουν αποσταλεί και θα θέλαμε να τα μελετήσετε γιατί είναι πολύ σοβαρή και ανησυχητική κατάσταση. Και σας παρακαλώ κυρίες και κύριοι να κρατήσετε ανοιχτή αυτή την έκθεση ώστε να μπορέσουν να, να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες αυτές για τις παραβιάσεις γιατί για αυτές τις τέσσερις παραβιάσεις δεν έχει δοθεί καμία απάντηση. Υπάρχουν όμως οι παραβιάσεις αυτές και θέλουμε να τύχει συνέχεια και να μην είναι ανοιχτή αυτή η αναφορά. Η ύπαρξη πολλών ζώων εξαρτάται από αυτή τη δράση σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Κατανοώ ότι για αυτές τις δύο αναφορές Υπάρχει ένα αίτημα διαφορετικό με την προηγούμενη. Η 1771 ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τροποποιήσει το νομικό καθεστώς των λύκων και να προστατεύσει πλήρως τους λύκους στην Ισπανία. Αν συγκρίνουμε τις δύο καταστάσεις, την Γερμανία και την Ισπανία, όπως είπα στη Γερμανία έχουμε ένα μικρό πληθυσμό από τα επίσημα στοιχεία που αναφέρονται στο 2007 με 12 μιλάμε 40 με 50 λύκους. Ίσως να έχει υπάρξει μια μικρή αύξηση πρόσφατα. Αλλά μιλάμε για μια, ένα πολύ μικρό πληθυσμό. Στην Ισπανία μιλάμε για χιλιάδες, χιλιάδες λύκους στη Γερμανία το νομικό καθεστώς είναι αυστηρά προστασία. Φόνος ενός, ε, η θανάτωση καλύτερα, ενός λύκου μπορεί να υπάρξει μόνο με ειδική άδεια ε, κατ' εξαίρεση. Στην περίπτωση στα βόρεια του Ντουέρο η νομοθεσία επιτρέπει ε, την θανάτωση των λύκων διαφορετικές συνθήκες σε διαφορετικές προβλέψεις και νομικά καθεστώτα. Ακόμα και η ευνοϊκή αυτή δημογραφική κατάσταση του ισπανικού πληθυσμού λύκων έχει επιβεβαιωθεί από την αξιολόγηση της ισπανικής κυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 17 της οδηγίας Χάμπιτας. Η αξιολόγηση αυτή έχει επιβεβαιώσει το καθεστώς ευνοϊκής ε, ε, επιβίωσης για τους λύκους και στην περιοχή του Ατλαντικού και στην ενδοχώρα. Κάποια αριθμοί που μας δίδουν για το μεσογειακό κομμάτι οι Ισπανικές αρχές αναφέρονται σε 1.200 με 1.800. Για το Ατλαντικό κομμάτι 650 ε, κεφαλές με χίλιες. Μιλάμε δηλαδή εδώ για μεγάλους πληθυσμούς οι οποίοι όπως είπα σύμφωνα με την οδηγία μπορούν να κυνηγηθούν εφόσον διατηρηθεί ο χαρακτηρισμός των λύκων ως έχει. Σύμφωνα με τις πληροφορίες τις οποίες έχουμε λάβει δεν εντοπίσαμε εμείς οποιαδήποτε παραβίαση της οδηγίας Χάμπιτας ε, για τη διαχείριση των λύκων από τις Ισπανικές αρχές. Τώρα για την ε, δεύτερη αναφορά. Οι άδειε κυνηγιού. Κατανοούμε ότι οι άδειε κυνηγιού ε, κατέστησαν διαθέσιμες μετά από αίτημα των ενδιαφερομένων δεν βλέπουμε να υπάρχει εδώ παραβίαση της ε, οδηγίας αυτής για την πρόσβαση σε περιβαλλοντικές πληροφορίες. Ε, η θανάτωση των λύκων στην περιοχή της Αστούριας δεν προϋποθέτει εξαίρεση σύμφωνα με το άρθρο 16 γιατί οι λύκοι στην συγκεκριμένη ε, κατηγορία, ανήκουν στην κατηγορία του παρατήματος 5 ως εκ τούτου δεν υπάρχει ανάγκη για τις Ισπανικές αρχές να αποδείξουν την ανυπαρξία εναλλακτικής λύσης και δεν υπάρχει ανάγκη να αναφέρονται σε διετή βάση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την συγκεκριμένη ρύθμιση, γιατί αυτό είναι κάτι που βρίσκεται εκτός της κατεξαίρεσης χορήγησης αδείας. Υπάρχει ένα πρόγραμμα στην Αστούρια από το 2002 και εγκρίθηκε ένα νέο στις 15 Μαρτίου του 2015. Ο αριθμός των μέτρων συντήρησης έχουν σαν στόχο να συνεισφέρουν στην διατήρηση της ιδιότητας αυτού του καθεστώτος, ευνοϊκή συντήρηση του είδους δηλαδή, και επίσης το Natura 2000 σε σχέση με την προθεσμία την εξαετή για τον καθορισμό περιοχών σαν ειδικέ περιοχές συντήρησης του είδους και λήψης κατάλληλων μέτρων. Στην περίπτωση αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει μια διαδικασία επί παραβάση. Έστειλε μια επιστολή προειδοποίησης τον Φεβρουάριο μήνα για παράβαση του άρθρου 4 παραγράφου 4 και του άρθρου 6 παράγραφος 1 της οδηγίας Άμπιτας. Πρόκειται για μια οριζόντια περίπτωση, δεν αφορά αποκλειστικά τους λύκους. Of community importance that were not... Αφορά την Ισπανική Πανίδα και τους χώρους, τις περιοχές για τις οποίες δεν ισχύει η προθεσμία των 6 ετών συνειδητοποιούμε ότι υπάρχουν κάποια νέα στοιχεία τα οποία ελήφθησαν πριν λίγες μέρες και δεν μπορέσαμε να τα αξιολογήσουμε μέχρι σήμερα όμως. Επί τη βάση των πληροφοριών που έχουμε στη διάθεσή μας λοιπόν δεν διαπιστώνουμε παραβίαση της νομοθεσίας χάμπιτας για τους λύκους της οδηγίας Habitat για τους λύκους. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν προβλέπεται να αλλάξει την ε, νομοθεσία και να αλλάξει τα παραρτήματα. Να πω επίσης όμως ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην παρούσα φάση ολοκληρώνει μια συνολική αξιολόγηση των δύο οδηγιών Natura και της Χάμπιτα και της λεγόμενης fitness. Ολοκληρώνουμε το fitness check Λειτουργία της οργίας δηλαδή. Την επόμενη εβδομάδα θα παρουσιάσουμε τα προκαταρκτικά ευρήματα αυτής της έρευνας. Προς στιγμή λοιπόν εμείς αξιολογούμε τον τρόπο με τον οποίο οι οδηγίες αυτές έχουν εφαρμοστεί μέχρι σήμερα και δεν προβλέπουμε στην παρούσα φάση να προχωρήσουμε σε ιεσδήποτε αλλαγές. Ένα τελικό σχόλιο τώρα για τη σημασία που έχει ο διάλογος ανάμεσα στους εμπλεκομένους. Θα πρέπει να μειωθούν τα επίπεδα σύγκρουσης ανάμεσα σε διαφορετικές ομάδες ανθρώπων, κυνηγούς, οργανώσεις προστασίας και κυβερνητικές δομές. Η μακροπρόθεσμη προστασία των λύκων και γενικότερα των θηρευτών απαιτεί την αποδοχή των μέτρων αυτών από το κοινό. Έχει σημασία λοιπόν να λάβουμε υπόψη όσο μπορούμε περισσότερο τα συμφέροντα όλων των εμπλεκομένων ομάδων. Προς την κατεύθυνση αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημιουργήσει μια πλατφόρμα για την συνύπαρξη των μεγάλων θηρευτών και των ανθρώπων. Δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2014 με τους ε, εκπροσώπους σε ευρωπαϊκό επίπεδο των ιδιοκτητών γεών, κυνηγών, ε, εκπροσώπων ε, και των ομάδων προστασίας ταράμβων κτλ. Στόχος είναι να προωθήσουμε το διάλογο και να ανταλλάξουμε πληροφορίες έτσι ώστε να υπάρξει αμοιβαία κατανόηση και να προωθήσουμε όσο μπορούμε περισσότερο κοινώ συμπεφωνημένες λύσεις ε, για αυτές τις καταστάσεις συγκρούσεων οι οποίες ε, για μας αποτελούν ένα πάρα πολύ μεγάλο κίνδυνο για την επιβίωση των μεγάλων θηρευτών. Σας ευχαριστώ. Οι συνάδελφοι έχουν τον λόγο. Πρώτη η κυρία Εύη. Ευχαριστώ να μου επιτρέψετε να σχολιάσω λίγο αυτές τις δύο αναφορές και σε σχέση με την προηγούμενη αναφορά. Στην Επιτροπή Περιβάλλοντος αυτή την εβδομάδα κάναμε ε, μία συζήτηση για την μεσοπρόθεσμη στρατηγική για την βιοπικιλότητα. Όλοι οι συνάδελφοι συμφώνησαν ότι η φύση αυτή τη στιγμή ε, ζητάει βοήθεια. Και εδώ θα συμφωνήσω με τα κίνητρα των αναφερομένων έτσι και αλλιώ ε, ε, και οι γενικότερες, οι ευρύτερες ε, ομάδες που ασχολούνται με τα θέματα της βιοπικιλότητας ζητούν να υπάρξουν μέτρα για την διατήρησή της. Σαν παράδειγμα ο τρόπος χρήσης των γεών είναι ένα πρόβλημα, συνεχώς υπάρχει η διεύρυνση των αστικών περιοχών και τσιμεντοποίηση ε, τμήματων της υπαίθρου. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη για την αξιολόγηση της κατάστασης των οικοσυστημάτων και της βιοπικιλότητας. Έχουμε λοιπόν εδώ μπροστά μας τώρα μια περίπτωση, θα έλεγα μια κατάσταση που συνδέεται με αυτό το θέμα Νομίζω ότι ακούσαμε κάποια θετικά στοιχεία. Ακούσαμε ότι κάθε πλαίσιο ξεχωριστό έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά. Οι αριθμοί των ζώων είναι εντελώς διαφορετικοί. Και να υπογραμμίσω επίσης ότι είμαι πεπισμένη για την ανάγκη η οποία υπάρχει να δραστηριοποιηθούμε εκ νέου στα πλαίσια του διαλόγου αυτού ανάμεσα στους γεωργούς από τη μία που είναι μια ομάδα πληθυσμού που θέλει να προστατεύσει τους αριθμούς των ζώων Εγώ είμαι βέβαια πεπισμένη ότι το κυνήγι είναι μια σκληρή και απαράδεκτη και βίαιη πρακτική και θα πρέπει ακριβώς να βρούμε διαφορετικά μέτρα για να προστατεύσουμε τα άγρια ζώα στην Ευρώπη. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα, πάρα πολλά μέσα τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και έτσι θα μπορέσουμε να σταθμίσουμε τα μεγέθη των αγρίων ζώων. Χρειάζεται περισσότερη προσοχή γιατί επαναλαμβάνω ότι η φύση ζητάει βοήθεια και δεν μπορούμε να πούμε ότι προστατεύουμε τη φύση. Γιάρεκ. Ευχαριστώ πολύ. Από νομικής απόψεως δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε η Επιτροπή μας ε, δεν έχει καμία δουλειά να ασχοληθεί περαιτέρω με αυτή την Επιτροπή. Προτείνω να την κλείσω. Δεν θέλω να είμαι όμως, ε, απλώς ας λάβουμε υπόψη ε, τα στοιχεία. Η οδηγία περί οικοσυστημάτων δεν έχει παραβιαστεί. Το κυνήγι εκεί είναι νόμιμο. Οι κυνηγοί λαμβάνουν άδειες προκειμένου να κυνηγήσουν. Και λαμβανομένων υπόψη όλων αυτών των στοιχείων, νομίζω ότι όλα είναι μια χαρά και όλα όσο συμβαίνουν εκεί ε, είναι νόμιμα. Οπότε δεν βλέπω τι μπορούμε να κάνουμε ως Επιτροπή. Προτείνω να κλείσουμε αυτές τις αναφορές. Mrs. Yes, Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ε, αναφέροντες ε, για την εργασία τους και δεν θα επαναλαμβάνω την έκκλησή μου για καλύτερη προστασία των λύκων. Ε, το έκανα στην προηγούμενη αναφορά. Δύο σημεία νομίζω μας, θα έπρεπε να μας οδηγήσουν στο να κρατήσουμε ανοιχτή αυτή την αναφορά το θέμα που έθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ε, τα ε, δεδομένα των ζώων που φανατώνονται. Γιατί δεν είμαι πάρα πολύ πεπισμένη ότι είναι τόσο διαφορετική η κατάσταση στην Ισπανία από ό,τι στη Γερμανία. Ε, το κυνήγι είναι σημαντικό και μεγάλης κλίμακας, οπότε θα ήθελα να επαναλάβω ότι είναι σημαντικό και πάλι να έχουμε καλά δεδομένα και να υπάρχει επιστημονική παρακολούθηση και ε, αναφορά των δεδομένων αυτών. Μία συμβουλή θα ήθελα να δώσω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά στο διάλογο. Όταν αρχίζεται ένα διάλογο για ε, καταστάσεις ε, επίμαχες να θυμάστε ένα πράγμα. Μην ξεχνάτε να δείτε και την άποψη των λύκων, γιατί στην απάντησή σας για την προηγούμενη αναφορά είπατε ότι ε, είναι φυσιολογική διαδικασία το να είναι ε, λία τα άγρια ε, ζώα για τους λύκους από ότι το να τρώνε οι λύκοι τα πρόβατα. Όμως άμα δείτε από την άποψη των λύκων την κατάσταση είναι φυσιολογική συμπεριφορά και η φύση τους και στις δύο περιπτώσεις. ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν Α, κυρία Βαλέρο. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε καλύτερες πληροφορίες σε σχέση με το επίπεδο θανάτωσης των λύκων στην Ισπανία. Πόσοι υπάρχουν και πόσοι θανατώνονται. Μας λένε πάνω από χίλιοι, αλλά ποια είναι η αναλογία κατέτος ε, της θανάτωσης. Αυτό είναι σημαντικό. Νομίζω ότι θα πρέπει να ολοκληρώσουμε για την αναφορά αυτή. Η πρότασή μου είναι η εξή. Άκουσα την άποψη του κυρίου ε, Βαλέσαν να κλείσουμε όλες τις αναφορές. Εγώ προτείνω για την πρώτη αναφορά 1771 να στείλουμε την ε, αναφορά στις ισπανικές αρχές ενημερωτικά για να ξέρουν ότι έχουμε εξετάσει το θέμα αυτό και μετά μπορούμε να την κλείσουμε. Όσον αφορά τώρα τη δεύτερη, νομίζω ότι οι νέες πληροφορίες τις οποίες λάβαμε τις τελευταίες ε, ημέρες πρέπει να αναλυθούν πλήρως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γι' αυτό προτείνω να παραμείνει ανοιχτή μέχρι να έχει χρόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να, ολοκληρώσει την ανάλυση των στοιχείων αυτών ενδεχομένως να λάβουμε και νέες πληροφορίες από αυτού. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Ποιος θέλει να πάρει το λόγο. Κυρία Χάουζερκαμπ. Ναι, κοιτάξτε. Υπάρχει τόσο μεγάλη διαφορά μεταξύ των δύο αυτών αναφορών. Εγώ δεν το βλέπω Αν δεν υπάρχουν μεγάλε διαφορέ, νομίζω ότι μπορούμε να τι κρατήσουμε και τι δύο ανοιχτέ μέχρι να γίνει ανάλογη, ε, ανάλυση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ναι, αλλά αυτό δεν έχει πολύ νόημα, λέει η Πρόεδρο, γιατί έχει γίνει πλήρη ανάλυση τη πρώτη αναφορά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μπορεί να κάνει σαφή αξιολόγηση και να πει ότι δεν γίνεται παραβίαση των διατάξεων τη οδηγία ε, οικοσυστημάτων, που ήταν ε, το θέμα τη αναφορά. Μπορεί να είστε συναισθηματικά φορτισμένοι ω προ αυτό. Από νομική απόψεω όμως τα πράγματα είναι διαφορετικά. Για τη δεύτερη αναφορά έχουμε περισσότερες πληροφορίες καινούριε που πρέπει να αναλυθούν. Γι' αυτό προτείνω ε, να πράξουμε όπως σα είπα. Κυρία Βαλέρο. Στα πλαίσια της πρώτης ε, αναφοράς έγινε μια παραπομπή σε, μια συγκεκριμένη, σε ένα συγκεκριμένο από τα παρατήματα. Πώς ακριβώς, ποια ήταν αυτή η παραπομπή. The information here. Οι πληροφορίες είναι ότι ποτέ δεν μας ε, δόθηκαν παραρτήματα, οπότε η θέση μας πρέπει να βασιστεί στις πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας. Γι' αυτό ακριβώς επανεπισημένω την πρότασή μου να κλείσουμε την πρώτη αναφορά και να αναλύσουμε πλήρως τη δεύτερη. Εντάξει, ωραία. Αυτό θα κάνουμε και τώρα πρέπει να προχωρήσουμε στη τελευταία αναφορά Έχουμε ακόμη 12 λεπτά, όμως ε, δεν είναι εδώ αναφέρον. Ε, σουηδική ενεφορά αναφορά αυτή. Σπάνιο Η φαινόμενο, ε, υπαριθμό 0011-2015 για τις ενέργειες τις οποίες προέβη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε υπόθεση που αφορούσε κυνήγι λύκων στη Σουηδία. Να σας εξηγήσω τώρα πώς έχει η κατάσταση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε διαδικασία επιπαραβάση κατά της Σουηδίας το 2010 σε σχέση με τη χορήγηση αδειών κυνηγιού και τον τρόπο με τον οποίο ε, εφαρμόζονται. Τον Ιούλιο του 2014 ξεκίνησε ε, διαδικασία δεύτερη φορά. Αυτή τη φορά το θέμα ήταν η πρόσβαση στη δικαιοσύνη και συγκεκριμένα η δικαστική αναθεώρηση των διοικητικών αποφάσεων που είχαν να κάνουν με τις άδειε κυνηγιού. Να δώσω τώρα το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας παρακαλώ να είστε όσο το δυνατόν πιο σύντομοι, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο σύντομη γίνεται. Η αναφορά στη συγκεκριμένη περίπτωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πράγματι χρειάστηκε χρόνο στα πλαίσια της διαχείρισης του θέματος των λύκων. Εμείς χρησιμοποιήσαμε την αρχή της επικουρικότητας από τη μία όπως προβλέπει η συνθήκη και την διακριτική ευχέρεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, να χρησιμοποιήσει μη την διαδικασία επί παραβάση. Εμείς θεωρούμε ότι η Εθνική Δικαστική Τάξη είναι καταρχάς υπεύθυνη για τις διαδικασίες αυτές και θα πρέπει να διασφαλιστεί πρώτα απ' όλα η προσφυγή στη δικαιοσύνη. Ε, στόχος αυτής της διαδικασίας είναι να δώσουμε στα κράτη-μέλη την δυνατότητα να εξηγήσει τις θέσεις της και μόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει την δυνατότητα να παραπέμψει τα κράτη-μέλη στο δικαστήριο. Η Σουηδία αποφάσισε στην αδειοδότηση θανάτωσης ε, λύκων από το 2011 και το συνέχισε το 2013, το 2014 και το 2015. Όπως είπαμε ξεκινήσαμε εμείς τις διαδικασίες επί το 2011 ήδη αποστέλλοντας δύο προειδοποιήσεις προς τη Σουηδία γύρω από το θέμα αυτό, το 13 και το 14, τα σουηδικά δικαστήρια ε, ασχολήθηκαν με το θέμα, υπήρχε δυνατότητα ε, του να εφεσιβάλει κανείς τις αποφάσεις αλλά συνεχίζονται οι ε, δραστηριότητες, οπότε σε αυτή την περίπτωση εμείς είπαμε ότι εφόσον ασχολούνται τα δικαστήρια δεν χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εμπλακεί. Το 2014 όμως άλλαξε το θέμα και η απόφαση από πλευράς της Κεντρικής ε, Υπηρεσίας Προστασίας Περιβάλλοντος ε, δόθηκε η δυνατότητα λήψης των αποφάσεων για την αδειοδότηση μη στις περιφερειακές, στα περιφερειακά συμβούλια. Και γι' αυτό ξεκινήσαμε μία δεύτερη διαδικασία προσφυγής επί παραβάσης βάρος της Σουηδίας τον Ιούλιο του 2014. Τον Οκτώβριο του 2015 οι Σουηδικές Αρχές δημοσίευσαν μία έκθεση σχετικά με τις εφέσεις οι οποίες έχουν γίνει σε σχέση με την αδειοδότηση κυνηγίου των μεγάλων θηρευτών. Εμείς θεωρήσαμε ότι αυτές οι ρυθμίσεις που ισχύουν σήμερα πρέπει να αλλάξουν γιατί είναι ασύμβατες με την κοινωνική ε, ένωμη τάξη και θα πρέπει να αλλάξουν το σύστημα το οποίο χρησιμοποιούν. Πάντως, σε σχέση με την προσφυγή επί παραβάση για την αδειοδότηση του κυνηγίου. Τρεις μεγάλες περιφέρειες αποφάσισαν το 2015 ε, να εκδώσουν 44 άδειε. Υπήρξε μια συμπληρωματική προειδοποίηση από πλευράς μας και χθες μόνο πέντε περιφέρειες αποφάσισαν εκ νέου από τις 16 Ιανουαρίου να επιτρέψουν το κυνήγι των λύκων για 46 λύκους. Εμείς μελετάμε το περιεχόμενο των προγραμμάτων αυτών. Έχουμε λοιπόν δύο διαδικασίες επί παραλήψη ανοιχτές σε σχέση με τη διαχείριση των λύκων και το κυνήγι των λύκων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του ρόλου που τους αποδίδουν οι συνθήκες έχει λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα τα οποία απαιτούνται στη συγκεκριμένη περίπτωση. Σας ευχαριστώ. Γιάρεκ, έχει το λόγο. Νομίζω ότι η κατάσταση εδώ είναι αρκετά απλή. Οι διαδικασίες επί παραβάση έχουν ξεκινήσει και θα πρέπει να κρατήσουμε τις δύο, την αναφορά αυτή ανοιχτή. Πράγματι έχει μεγάλο ενδιαφέρον ε, για τον υπόλοιπο κόσμο η κακή συμπεριφορά της Σουηδίας στο συγκεκριμένο τομέα. Δεβαλέρο. θα ήθελα να μιλήσουμε, ε, ε, πράγματι προκαλεί πάρα πολύ ενδιαφέρον η συζήτηση αυτή και θα θέλαμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δράσει στις περιπτώσεις αυτές ακόμα πιο γρήγορα από όσο το κάνει. Αυτό θα μας βοηθήσει για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε το είδος αυτό. Λοιπόν, μπορούμε να το κλείσουμε αυτό. Ε, υπάρχουν δύο, παραβάσεις, δύο διαδικασίες επί παραβάσεις βάρος της Σουηδίας. Χρειάζεται λοιπόν να κρατηθεί ανοιχτή η διαδικασία Ελπίζω οι πράσινοι να μας ακούσουν λίγο, να κάνουν λίγη ησυχία. Νομίζω ότι τα συμπεράσματα λοιπόν από τη συζήτηση αυτή ε, θα βοηθήσουν την διατήρηση των λύκων και τη διαχείριση ε, του προβλήματος. Υπάρχουν δύο διαδικασίες λοιπόν ανοιχτές και κρατάμε τις αναφορές αυτές γιατί σε οριζόντιο επίπεδο ε, εμείς θα αντιμετωπίσουμε με τον ίδιο τρόπο και τις επόμενες ε, αναφορές ε, ανεξαρτήτως ε, της πλευράς από την οποία προέρχονται. Σε επίπεδο νομικό κρατάμε ανοιχτές γιατί πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε σύμφωνα με, με την κατάσταση οποία νομική η οποία ισχύει. Λοιπόν η οδηγία αυτή παραμένει ανοιχτή και αυτό εξυπηρετεί συνολικότερα το συμφέρον του σώματος αυτού που είναι να παρακολουθήσει από κοντά την διαδικασία της διαχείρισης των λύκων στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Υπήρου. Λοιπόν, συμφωνείτε? Εντάξει, σας ευχαριστώ. Αυτό ήταν το τελευταίο θέμα για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για μια πολύ ενδιαφέρουσα και καρποφόρο συνεργασία. Σας εύχομαι καλό απόγευμα.